Ladies and Κυρίες και κύριοι, σας παρακαλώ καθίστε. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην απογευματινή αυτή συνεδρίαση της Υποεπιτροπής ε, Ασφάλειας και Άμυνας. Ως συνήθως θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ε, μεταδίδεται διαδικτυακά η συνάντηση, η συνεδρίαση αυτή και ο συνήθως ε, δίνεται προτεραιότητα στη διερμηνία στις γλώσσες των πλήρων μελών της Επιτροπής ε, Άμυνας και Ασφάλειας. Δεν έχουμε να εγκρίνουμε πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων, διότι έχουν ήδη εγκριθεί. θα έχουν, α, μάλλον θα τα υποβάλουμε στο πρώτο 15 του Οκτωβρίου ε, τα πρακτικά αυτή τη συνεδρία τη Υποεπιτροπή και θα ήθελα τώρα να περάσω απευθεία στην έγκριση τη ημερήσια διάταξη. Η γραμματεία με ενημέρωσε ότι υποβλήθηκαν ερωτήσεις και έγιναν σχόλια από πολιτικές ομάδες όσον αφορά το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, τη συνεδρίαση για την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή που θα παρουσιαστεί από τη Σκοπιά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Θέλω να σας ενημερώσω ότι πρόκειται για την πρώτη από μια σειρά παρουσιάζων επί του θέματος. Θεωρούμε ότι το θέμα αυτό θα είναι σημαντικό στο επόμενο διάστημα. Αποφασίσαμε να ακούσουμε τις αμερικανικές και ισραηλινές απόψεις εν ώψη ε, της ε, κοινή επίσκεψης ΑΦΕΤ και της Επιτροπής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες τον ερχόμενο μήνα, θέλαμε να ακούσουμε τις θέσεις ε, των Αμερικανών για θέμα, στο θέμα της ε, κατάστασης ασφαλείας στη Μέση Ανατολή. Και κατόπιν θα προσπαθήσουμε πριν την κοινή ad hoc αποστολή να κανονίσουμε, να γίνει συνάντηση επί του, πάνω κάτω επί του ιδίου θέματος, όπου θα παρουσιαστούν οι επίσημες ε, απόψεις της ε, EAS και των διαφόρων think tank των Βρυξελών, της υπηρεσία εξωτερικής, της ε, εξωτερική... Αλλά δυστυχώς έγιναν ε, αλλαγές, εσωτερικές αλλαγές στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης και ο, πιο αρμόδιος, ο διευθυντής κύριος Ουμπράλ, ε, ε, ανώτατος τέλεχος της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, άλλαξε αρμοδιότητες και ως εκ τούτου δεν έχουμε κάποιον και πιστεύουμε ότι πρέπει να περιμένουμε λίγο ώστε να καλέσουμε ε, κάποιον που θα είναι πλέον έτοιμος να παρουσιάσει τις επίσημες θέσεις της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. ήταν απόφαση των ε, θεσμική να γίνει αυτή η αναβολή. Ε, θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε τις θέσεις της Επιστροπής της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης το ταχύτερο δυνατόν. Ελπίζω πριν ε, να αναχωρήσουμε για Νόρφολ και Ουάσιγκτον τις παρατηρήσεις αυτές. Ελπίζω να είσαστε έτοιμοι και διατεθειμένοι να ε, εγκρίνετε την ημερήσια διάδεξη. Κύριε Γκάλερ, το σημειώνω αυτό, Πρόεδρε. Παρά τα αυτά, θα ήθελα να είχε γίνει συζήτηση γιατί ο τρόπος που συνήθως χειριζόμαστε τα πράγματα είναι να παρίστανται και τα θεσμικά όργανα όταν, ε, τα θεσμικά μας όργανα όταν έχουμε ε, επισκέπτες ε, τρίτους. Θα ήθελα αυτό να συνεχιστεί στο μέλλον. Πρόεδρος, βεβαίως ε, ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι προσπαθήσαμε, απλώς η κατάσταση αυτή οφείλεται στις αλλαγές εντός της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης και προσπάθησα να πω σαφώς ότι επιδιώκουμε να ακουστεί η άποψη των ΗΠΑ και του Ισραήλ αυτή τη στιγμή και ότι σκοπεύουμε ε, να συνεχιστεί η σειρά των ε, συναντήσεων. Ευχαριστώ για την παρατηρήσή σας. Ελπίζω ότι τώρα εγκρίνεται η μερίσια διάταξη και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση θα περάσω στο πρώτο θέμα της μερίσιας διάταξης και να καλωσορίσω θερμά τον ε, επισκέπτη που έρχεται εδώ συχνά. Έχουμε την τύχη να έχουμε μαζί μας τον κύριο Χόρχερ Ντόμεκ που είναι εκτελεστικός διευθυντής ε, του, Ευρωπαϊκής... Ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Σήμερα θα μας ε, μιλήσει για, τον... για την μακροχρόνια μακροπρόθεσμη αναθεώρηση του οργανισμού. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής ε, που μου δίνετε την ευκαιρία για μία ακόμα φορά να απαντήσω, να απευθυνθώ στην Υποεπιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδίως η Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι δίνει μια όθηση στις καινοτόμες ε, ε, προτάσεις. Θα ήθελα εδώ να υπενθυμίσω την ιδέα του πιλωτικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έρευνα σε σχέση με τον χώρο της άμυνας που προήλθε από αυτή την Επιτροπή και που τώρα υλοποιείται από τον οργανισμό. Θα επανέλθω σε αυτό στην επόμενη συνεδρία. Είμαι πεπισμένος ότι το Κοινοβούλιο θα μπορέσει να δώσει περαιτέρω όθηση τα επόμενα μήνες και τα χρόνια ε, οπωσδήποτε είναι εντάσσεται στις συστάσεις και τις γνωμοδοτήσεις που έχουν δημιουργηθεί, ε, προκύψει από αυτό το χώρο. Και για τον λόγο αυτό είμαι ιδιαίτερο ευγνώμων που είμαι σε θέση να συζητήσω ε, μαζί σας την λεγόμενη μακροπρόσφυνα θεώρηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, του LTR με δύο ε, συντομία. Θα ήθελα να σας, πει, ε, να σας πω ευθύ εξ αρχή ότι ο LTR είναι βασική προσπάθεια και ένα σημείο καμπή για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα. Έχει ενισχύσει την αποστολή του οργανισμού και έχει προωθήσει τι φιλοδοξίε απέναντι στο ρόλο του οργανισμού σε σχέση με, την, με τις διάφορες ε, υποεξέλιξη πρωτοβουλίες όπω είναι ΠΕΣΚΟ, ΚΑΡΔ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. Η διαδικασία LTR ξεκίνησε από την επικεφαλής της υπηρεσίας, τη Φεντερίκα Μοκερίνη και ο σκοπός είναι να μπορέσει να, είναι, να ανταποκρίνεται στο σκοπό της και να έχει επαρκή μέσα ε, ε, πάνω από 12 χρόνια αφότου πρώτο δημιουργήθηκε. Η προσπάθεια της ε, μακρο πρόθεσμης αναθεώρηση αποτελείται από μια σειρά υψηλού επίπεδου συναντήσεων που πραγματοποιούνται στο εξάμεινο Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν στο εξάμεινο Νοεμβρίου Απριλίου 2017, ε, κατά, ε, κατά τις οποίες έγινε ε, ε, εξέταση σε βάθο και μια διαρθρωμένη αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων στόχων του Οργανισμού Άμυνα. Ε, ποια είναι τα βασικά σημεία που εντοπίστηκαν. Η μακροπρόθεσμη αναθεώρηση υποστηρίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν τρεις βασικές λειτουργίες του Οργανισμού Άμυνας. Πρώτον, να λειτουργήσει ως το μέσο, το βασικό μέσο, το οποίο θα θέτει προτεραιότητες διακυβερνητικά. Ε, ανάμεσα στην ε, Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και τη Στρατιωτική Επιτροπή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θέση προ... Ε, προτεραιοτήτων είναι το βασικό όρο εδώ. Αυτό σημαίνει η κατανόηση του τι είναι ε, διαθέσιμο και τι δεν είναι διαθέσιμο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να επικεντρωθούν οι πόροι προ αυτό το οποίο πραγματικά είναι απαραίτητο. Έχουμε το σχέδιο ανάπτυξη δυνατοτήτων, το λεγόμενο CDP, το οποίο προσδιορίζει ποιε δυνατότητε θα χρειαστούν για να εξυπηρετηθεί το γενικό επίπεδο φιλοδοξίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί να αναπτυχθεί σε συνεργασία ε, λαμβάνοντας υπόψη και την προσφορά των κρατών μελών στο ΝΑΤΟ. Το CDP επανεξετάζεται τώρα σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και οι νέε προτεραιότητες δυνατοτήτων αναμένεται να εγκριθούν μέχρι τον επόμενο Μάρτιο. Η σχέση με τα εθνικά σχέδια θα ε, ε, είναι όλο και πιο σημαντικά στην εξασφάλιση μιας ε, ε, συνεκτικής αποδοχής και της αποτελεσματικής υλοποίησης των συγκεκριμένων τομέων προτεραιοτήτων. Οι προτεραιότητες του CDP θα πρέπει επίσης να ενημερώνουν και να καθοδηγούν την μελλοντική ε, έρευνα στον τομέα της άμυνας που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας. Αυτό όσον αφορά την έρευνα και την τεχνολογία και τις σχετικές δραστηριότητες, αναπτύσσουμε περισσότερο το γενικό πρόγραμμα στρατηγικής έρευνας, έτσι ώστε να ενισχύσουμε τις στρατηγικές ε, προσπάθειες και να καταλήξουμε στις σωστές προτεραιότητες είμαστε ε, τελικά ε, στραμμένοι στο να εντοπίσουμε τις βασικές στρατηγικές δραστηριότητες, να εντοπίσουμε τις ε, βιομηχανικές δυνατότητες και δεξιότητες που χρειάζεται η Ευρώπη. Εντάσσουμε στο ενιαίο πλαίσιο αυτά τα εργαλεία για να υπάρχει μια γενική εικόνα σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές δυνατότητες και για την υλοποίηση βέβαια των προτεραιοτήτων μας στον τομέα CDP θα προσθεθεί στην εργαλειοθήκη και η συντονισμένη ετήσια αναθεώρηση της άμυνας, ε, κάτι το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει δοκιμαστικά. Και στόχο έχει ουσιαστικά να δώσει μια πλήρη εικόνα ε, του όλου τοπίου και της ε, υλοποίησης των δύο CDP. Μπορεί, βέβαια να έχετε ρωτήσει, οπότε μπορώ να επανέλθω αργότερα. Σε ό,τι αφορά τώρα την ΠΕΣΚΟ, τα κράτη-μέλη έχουν ζητήσει από τον οργανισμό σε στενή συνεργασία με το στρατιωτικό ΤΕΛ να υποστηρίξει μια, πρέτη, μια πρώτη ανάλυση των προτινόμενων έργων ΠΕΣΚΟ. Θα υπάρξει μάλιστα εργοστάς, εργοστήριο, συγγνώμη, workshop κατά τα τέλη Οκτωβρίου για το θέμα αυτό όπου θα παρουσιαστούν και τα πρώτα πορίσματα. Ο ρόλος του οργανισμού στην όλη διακυβέρνηση ΠΕΣΚΟ θα αναπτυχθεί τι επόμενε εβδομάδε επόμενου μήνε μήνες, σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν οι συνθήκε και οι διατάξει του Συμβουλίου και βέβαια λαμβάνοντα υπόψη τα πρόσφατα συμπεράσματα τη μακροπρόθεσμη αναθεώρηση. Χρειαζόμαστε φιλόδοξη ΠΕΣΚΟ που θα σημειώσει ποιοτικό άλμα σε ό,τι αφορά την αμυντική συνεργασία, είτε πρόκειται για ΚΑΡΤ, είτε για ΠΕΣΚΟ, είτε για CDP. Πιστεύουμε ότι η συμμετοχή ε, και η όθηση από τα κράτη-μέλη είναι κλειδιά επιτυχίας. Τώρα θέλω να στραφώ στη δεύτερη βασική λειτουργία που έχει αποδοθεί στον οργανισμό μας, ε, στο πλαίσιο της ε, μετακόρποτες μεσανθεώρησης. Ο οργανισμός θα πρέπει να είναι το προτιμητέο φόρουμ συνεργασίας και δομή υποστήριξης σε ό,τι αφορά την τεχνολογία και την ανάπτυξη δυνατοτήτων. Αυτό αναγνωρίζει ουσιαστικά το έργο του οργανισμού που εδώ και χρόνια επιτελεί. Ο οργανισμός συμμετέχει σε πολλές δραστηριότητες που προωθούν τη συνεργασία. Διευκολύνει το διάλογο μεταξύ κρατών μελών, καταρτίζει μελέτη κοπιμότητας για τον εντοπισμό περαιτέρω δυνητικά ε, περιοχών ή τομέων συνεργασίας και στηρίζει ή πολλών έργων και σχεδίων. 50 έργα στον τομέα των δυνατοτήτων και γύρω στα 100 στον τομέα τη Έρευνα και τεχνολογίας υποστηρίζουμε στο πλαίσιο του οργανισμού μας αυτή τη στιγμή. Σε ό,τι αφορά τι πρόσφατε πρωτοβουλίε από το Μάιο και μετά, που τονίζουν ε, τι δυνατότητε του οργανισμού μα για τη στήριξη των ε, αναπτύξεων δυνατοτήτων, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τον ε, την εγγενία στο European Tactical Airlift Center τον Ιούνιο του 2017. Την διάσταση Cyber είχαμε μια άσκηση Seabridge σε πολιτικό επίπεδο το Σεπτέμβριο. Επίσης ε, είχαμε την συγκρότηση μιας ad hoc ομάδας εργασίας για την στρατιωτική ε, μεταφορά το Σεπτέμβριο και έχουμε και άλλες πρωτοβουλίες που εξελίσσονται όπως το Main Battle Tank και πολλοί άλλοι τομεί υπάρχουν, στου οποίου θα μπορούσαμε να δώσουμε μια ευρωπαϊκή διάσταση στο μέλλον ω οργανισμό άμυνα. Τρίτο βασικό καθήκον προβλέπεται η ενίσχυση του ρόλου του οργανισμού μας ως ε, παράγοντα διευκόλυνσης προς την Κομισιόν και άλλους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Central Operator συγκεκριμένα, αυτός είναι ο ρόλος μας για τις δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την άμυνα και χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, που είναι ο σύνδεσμος αφενός μεταξύ των κρατών και αφετέρου μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Ο οργανισμός από θεσμικής πλευράς είναι ξεθέσει να διδραματίσει το ρόλο αυτό. Υπάγεται στο Συμβούλιο, ωφελείται και λαμβάνει άμεση πολιτική αυτοδιοίκηση από τους πλούς άμυνας, αλλά και άλλους, όπως είναι οι, διεθνοί, οι διευθυντές εθνικού εξοπλισμού, οι διευθυντές οι διευθυντές έργας τεχνολογίας, ή αμυντική πολιτική. Ένα από του βασικού στόχου μα είναι να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο ευρύτερων πολιτικών τη Ένωση, καθώ και κανονισμών, στον τομέα όπως ε, κυβερνοχώρο ε, διάστημα, ενέργεια. Ένα το παράδειγμα είναι ο ρόλο που έχει διδραματίσει από το 2010 ο οργανισμό στο συντονισμό των στρατηγικών απόψεων για το Single European Sky. Είναι μια διεπαφή διασύνδεση τη στρατιωτική κοινότητα με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και άλλου εταίρου, όπω είναι το Eurocontrol και το NATO. Τώρα, Έρχομαι στο ρόλο μας, όπως σας είπα, Central Operator για τις δραστηριότητες άμυνας που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεχίζονται οι συζητήσεις. Παράλληλα εφαρμόζουμε το πιλωτικό project και είμαστε και στο πρώτο έτος της προπαρασκευαστικής ενέργειας για την αμυντική έρευνα. Δεν έχει καθοριστό μας επαρκώς όρο Central Operator. Τι θα πει ακριβώς, ιδίως ό,τι αφορά το Capability Window και το EDITP, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής έχει δημιουργηθεί εντό τη υπηρεσία μα μια task force και τα κράτη-μέλη θα δώσουν τι απόψει του για το πώ ακριβώ θα βοηθήσει ο οργανισμό στα κράτη-μέλη. Έχουμε ήδη παράσχει συμβουλές ε, στο πλαίσιο των φίλων τη Προεδρία αυτή τη ομάδα του Συμβουλίου για το μέλλον τη συμμετοχή των ε, ΜΜΕ στα ΕΔΙΤΠ, στου ε, μελλοντικού διαγωνισμού. Και θα υπάρξει και ένα consultation forum στο οποίο θα δώσουμε πάλι τη γνώμη μας. Σε ό,τι αφορά τώρα το, τις προτάσεις ε, ΠΕΣΚΟ, αντίστοιχα θα μπορούσαμε να δίνουμε συμβουλές και για το EDITP σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ζητήσαμε και τη στήριξη των κρατών μελών αυτό δεν είναι παρά μια φυσική απόρρεια της ε, έκκλησης των κρατών μελών ε, να διασφαλιστεί η απαιτούμενη διασύνδεση μεταξύ ΚΑΡΤ, ΠΕΣΚΟ και EDF. Ναι, μεν είναι ξεχωριστές αυτές οι πρωτοβουλίες, αλλά όλες έχουν ως στόχο να βελτιώσουν την συνεκτικότητα του τοπίου δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα τι προτεραιότητες που έχουν συμφωνήσει. Να μην ξεχνάμε ότι τελικά το EDF, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας δηλαδή, δεν θα πρέπει να είναι απλά μια επιδότηση αλλά να οδηγήσει στην ανάπτυξη των απαιτούμενων δυνατοτήτων βάσει μιας ισχυρής ευρωπαϊκής αμυντικής, τεχνολογικής και μηχανικής βάσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει διασύνδεση με τις προτεραιότητες ε, και τη δημιουργία δυνατοτήτων και αυτό είναι ο ρόλος μας. Γι' αυτό και ο κανονισμός EDITP θα πρέπει να είναι κάτι που θα μας απασχολήσει και του σύνεγγις. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό επίσης είναι η σωστή ισορροπία μεταξύ της κοινοτικής και της διακυβερνητικής διάστασης. Αν θέλουμε βέβαια η αμυντική συνεργασία να σημειώσει ένα ποιοτικό άλμα. Κατά την αποψή μου, αυτό είναι το δομικό ζήτημα με δέλτα κεφαλαίο, επί το οποίο βασίζονται όλες οι επιτυχίες όλων των προσπαθειών μας. Τι θα πει σωστή ισορροπία. Θα πει ότι κάθε φορέας θα πρέπει να παίξει το ρόλο του. Θα συνάδει με τα καθήκοντα που έχει, την εντολή, την εμπειρία και τις αρμοδιότητες, ευθύνες. Θα πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση ρόλων, όπως προβλέπονται αυτοί από τη συνθήκη και από την πολιτική πραγματικότητα επιτόπου. Να μην ξεχνάμε ότι ο οργανισμός άμυνας αναφέρεται και στη συνθήκη ως οργανισμός που είναι αρμόδιος στον τομέα της ανάπτυξης αμυντικών δυνατοτήτων, της, α, της έρευνας, συγγνώμη, των α, δημοσίων προμηθείων και των εξοπλισμών. Θα ε, συνεχίσει δε η άμυνα, από ό,τι φαίνεται για το προβλεπόμενο μέλλον, να είναι ε, εθνική αρμοδιότητα. Το λέει και η συνθήκη, που σημαίνει ότι οποιοδήποτε σημαντικό βήμα προς την αμυντική συνεργασία θα γίνει πραγματικότητα μόνο αν συμμετέχουν ε, σε αυτή την προσπάθεια τα κράτη-μέλη ενεργά. Μπορούμε ως Ευρωπαϊκή να δώσουμε σημαντικά κίνητρα, αλλά και χρηματοδότηση. Γι' αυτό και χαιρετίζουμε την δημιουργία του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Ταμείου. Χρειάζεται όμως παραπάνω εξωτερικά ερθίσματα για την ενίσχυση της ε, συνεργασίας που δεν είναι αντανακλαστικό φυσικό. Δεν χρειάζεται όμως ταυτόχρονα αλληλεπικάλυψη δομών, γιατί αυτό σημαίνει απώλεια πόρων και σύγχυση στο, σε ό,τι έχει να κάνει με τις θεσμικές αρμοδιότητες. Πρώτα η πολιτική, μετά οι δομές και όχι ανάποδα. Θα πρέπει να αξιοποιηθεί λοιπόν πλήρω ο οργανισμός άμυνας, που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε και τους κατάλληλους και επαρκείς πόρους στη διάθεσή μας. Ε, μιλάω και για ανθρώπινους πόρους και για ε, οικονομικούς και για την ε, κατάλληλη λήψη αποφάσεων. Έγινε λόγος και για την ε, δυνητική αξία της ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία που το λέει και ε, η απόφαση του Συμβουλίου που θεσπίζει τον οργανισμό και αναγνωρίζεται εκεί επίσης ότι θα πρέπει ο οργανισμός να έχει τους απαιτούμενους πόρου και τα απαιτούμενα προγνωμοσύνη. Το κοινοβούλιο σας, θέλω να τονίσω εδώ, έχει και αυτό επιχειρηματολίσει πέντε της ενίσχυσης χρηματοδότησης και των μέσων του οργανισμού. Ένα άλλο θέμα το οποίο αντιμετωπίσαμε στη διάρκεια αυτής της ε, μακροπρόθεσμας ανθεώρησης ήταν οι αρχές που διέπουν τις σχέσεις μας με τρίτους. Μπορούμε να έχουμε σχέσεις με τρίτους, χώρες, οργανισμού ή άλλους φορείς για να φέρουμε σε πέρα στην αποστολή μας. Και το μόνο όχημα για την επίσημη συνεργασία είναι η σύναψη μιας ε, ε, διοικητική ρύθμιση, μιας, ενό διοικητικού διακανονισμού. Αφού ζητηθεί αυτό ρητό από τον ενδιαφερόμενο τρίτο και θα πρέπει βέβαια να εγκριθεί ομόφωνα από το Συμβούλιο. Έχουμε τέτοιε συμφωνίε με Νορβηγία, Ελβετία, Δημοκρατία Σερβία, Ουκρανία, όπω επίση με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και το ΟΚΑΡ. Αυτά που συζητήσαμε στη διαδικασία τη μακροπρόθεσμη μας με τα κράτη-μέλη ήταν οι αρχέ που θα διέπουν τι σχέσει ε, του οργανισμού με τρίτου. Συγκεκριμένα. Έχουμε σχέσεις και επαφές με τρίτες χώρες ε, σε πλήρη διαφάνεια με τα κράτη-μέλη. Όταν λαμβάνουμε τρεις παράγοντες, τρία πράγματα, την κοινή πολιτική ασφάλειας και εξωτερική πολιτική, στρατηγικές εταιρικές σχέσεις, δεύτερον, τις πολιτικές ευαισθησίες των κρατών και τρίτον, την ανάγκη να γίνει σεβαστή απόφαση μάλλον η αυτονομία του οργανισμού στις δικασίες λήψη αποφάσεων. Η συνεργασία δεν είναι ένας τρόπος υποστήριξη εταίρων, είναι μια αμοιβαία ισορροπημένη σχέση με κοινό στόχο, την ανάδειξη δυνατοτήτων μέσω συνεργασία. Αυτό μπορεί να εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα με τρίτε χώρε, ένοπλε δυνάμει που λαμβάνουν χώρε επιχειρήσει σε CSDP. Οι διοικητικέ αυτέ ρυθμίσει δεν μπορούν να είναι καινογράμμα. Οι τρίτοι έχουν ε, την ευθύνη να δείξουν ότι πραγματικά δεσμεύονται ότι θα ακολουθήσουν αυτές τις διαδικασίες, θα είναι συνεργάσιμες, ε, συνεργάσιμοι με τον οργανισμό και τα κράτη-μέλη. Και βέβαια υπάρχει πλήρης ευελιξία και σε κατά περίπτωση βάση εκτελήσονται οι δραστηριότητες. Βέβαια το πιο δύσκολο το έχουμε μπροστά μας και θέλω να πω εδώ ότι οι αμυντικοί φορείς είναι αυτοί που θα πρέπει να, να οικειοποιηθούν την όλη αυτή διαδικασία και να εφαρμόσουν τις πρωτοβουλίες όπως η PESCO, CAR, DDF. Και θα πρέπει λοιπόν να αναζωογονηθεί, να ενισχυθεί ακόμη περιττέρου ο οργανισμός ως διακυβερνητικό εργαλείο. Μπορεί να υπάρχουν αυτές οι μεμονωμένες δράσεις και τα τεχνικά μέτρα, αλλά αν θέλουμε να πετύχει θα πρέπει τα κράτη-μέλη να δείξουν πολιτική βούληση, να έχουν συνεργατικές προσπάθειες στο πλαίσιο του οργανισμού και να δώσουν προβολή στην προσθέμενη αξία σε ό,τι αφορά τι οικονομίε κλίμακα και την ανάπτυξη δυνατοτήτων. Και εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να βοηθήσει, δηλαδή να δώσει σε στην κατεύθυνση τη σταδιακή δημιουργία μια Ευρωπαϊκή Άμυνα πιο φιλόδοξη, αξιοποιώντα πλήρω τον οργανισμό και άλλε σχετικέ δομέ. Αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε πάνω στην υλοποίηση των πρακτικών μέτρων για να φέρουμε σε πέρα τόσο αποφασίστηκαν στην αναθεώρηση και την άνοιξη του 2019 οι υπουργοί θα κάνουν έναν απολογισμό της προόδου και θα δουν κατά πόσο χρειάζεται να υποβληθούν περαιτέρω συστάσεις και να γίνουν και άλλα ε, βήματα. Δεν είναι δηλαδή μια διαδικασία άπαξ, ε, κάποιες, αποφάσεις, κάποιες αποφάσεις που ελήφθησαν το LTR, είναι μια συνεχής διαδικασία για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση στρατηγικό επίπεδο και στις πρωτεύουσες ε, και περισσότερη οικειοποίηση από τα κράτη-μέλη. και, όπως λέει και η Παγκόσμια Στρατηγική, η πλήρης αξιοποίηση του δυναμικού του οργανισμού είναι ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα για τις προσπάθειες στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Ολοκληρώνω με αυτά και είμαι στη θέση να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Domek. Now... Σας ευχαριστώ κύριε Ντόμεκ. Ο κ. Γκάλερ πρώτος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ντόμεκ που ξανάρθατε. Άκουσα αυτά που είπατε ήχησαν ως μουσική στα ότα μου. Περιγράψατε δυνατότητες, ποικίλε. Τώρα χρειάζεται πολιτική βούληση, ούτως ώστε κάτι μέρη να χρησιμοποιήσουν πλήρως τα υπάρχοντα. Να χρησιμοποιήσουμε τις διατάξεις συνθήκης, να εργοποιήσουμε και την ΠΕΣΚΟ μέχρι το τέλος του έτους τη συνεργασία αυτή και να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε του, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αμήνης. Ευχαριστώ που μας ενημερώσατε για τη συμβουλευτική ομάδα. Ευχαριστούμε που αναφερθήκατε στη μακροπρόθεσμη αναθεώρηση. Είπατε ότι το Μάρτιο θα το συζητήσουν το θέμα οι Υπουργοί, θα δουν που βρισκόμαστε. Μετά βέβαια το θέμα που τίθεται η εφαρμογή όλων αυτών και ενεργοποίηση της ΠΕΣΚΟ. Κατά τα άλλα, ίσως θα θέλαμε περισσότερες λεπτομέρειες. Κάτι άλλο, ερώτηση. Μία από τις συστάσεις της διευθύνουσας ομάδας. Σε κάποια φάση είχαμε πει κάτι για τη χρηματοδότηση για τη στελέχωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αμήνη και κάποιο κόστο να βγαίνει από τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, κάτι που ενεκρίθη από το Διευθυντικό Συμβούλιο. Ετέθη ότι πρέπει να ελεγχθεί. Ξέρουμε ποια είναι η θέση των κρατών μελών σχετικά με αυτό. Αναφερθήκατε και στο CARD, την ετήσια αναθεώρηση των αμυντικών ζητημάτων. θα θέλαμε περισσότερες πληροφορίες. Τι ακριβώς έχουμε. Τα κράτη-μέλη, πώς το βλέπετε. Συμμορφώνονται. Θα μοιραστούν τα στοιχεία τους με τους άλλους εταίρους για να έχουμε μια καλή συνολική εικόνα, να ξέρουμε τι έχουμε και τι χρειαζόμαστε. Τέλος. Αναφερθήκαμε στο πιλωτικό πρόγραμμα. Είμαστε στην προπαρασκευαστική δράση για την αμυντική έρευνα. Περισσότερα στοιχεία έχετε. Ευχαριστώ κύριε Γκάλερ. Ο Γιάνν Πασκό θέλει να πάρει το λόγο. Είναι εδώ. Α, είναι, εδώ είναι. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Ενθαρρύνθηκα τα μάλα από τον αυξανόμενο ρόλο του οργανισμού. Όπως αναφέραμε προηγουμένως εδώ, είστε ο καλύτερος, η καλύτερη βάση για τη συνεργασία και για την αύξηση του ρυθμού συνεργασίας. Υποθέτω ότι όλες οι προσπάθειες θα δημιουργήσουν κλίμα εμπιστοσύνης, ούτως ώστε να συμμετέχουν όλοι και περισσότεροι χώρες, αυτό από τη μια, και από την άλλη θα δοθεί αναγκαία όθησης για συνεργασία στην ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επενούμε λοιπόν τη δραστηριότητά σας. Υποσχόμεθα ότι θα κρατήσουμε την επαφή μεταξύ μας και μπορείτε να βασιστείτε επάνω μας. Θα σας στηρίξουμε. Ευχαριστώ. Ο κ. Χαβιέρ Νάρτ έχει το λόγο. Εγώ τρέφω βαθύτατο σεβασμό προς τον οργανισμό. Ταυτόχρονα όμως και βαθύτατη απογοήτευση με διακατέχει. Μπορεί να είναι άξιο επένων το έργο σας. Το πρόβλημα είναι η λογική. Δεν είναι καλό ή κακό. Είναι αναπόφευκτο να υπάρχει. Έχουμε τους πολιτικούς και μηχανικούς λόγους που δίνουν την απάντηση κάθε χώρα που κατασκευάζει όπλα έχει τη δική της πολιτική εξοπλισμών σε σχέση και με το σύστημα έρευνα και τεχνολογίας, ε, εμπορίας και πολιτικής τοποθέτησης. Έχουμε τη Βρετανία, ακόμη μέλος της Ένωσης, που πουλάει όπλα σχεδόν μπορώ να πω γελώντας και χλεβάζοντας τις οκτώ ε, τα κριτήρια που υπάρχουν και, λαμβάνει υπόψη ε, μόνο τα δικά της φέρντου. Θα πρέπει να υπάρχει τυποποίηση και διαλειτουργικότητα των συστημάτων. Είναι προφανές. Το ξέρει και ο, ο κάθε δεκανέας σε κάθε χώρα ότι στην οπισθοφυλακή κερδίζεται ο πόλεμος με την επιμελητεία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αν το πολυπλασιάσουμε αυτό με 100 και πάνω συστήματα, αυτό είναι πραγματικά για γέλια. να αστείο. Και τα στρατιωτική απειλή που δεν νομίζω ότι υπάρχει εγώ, αλλά τέλο πάντων η Ρωσία και κάτι άλλο. Επιθύρας έχουμε την σύγκρουση στα ανατολικά και εσωτερικά έχουμε το Σαχέλ. ξύπνησαν τα κράτη-μέλη, αφυπνίστηκαν με όλες αυτές τις κρίσεις. Και εκτός από το Ραφάλ, το Γαλλικό και άλλα Βρετανικά και τα λοιπά, σκέφτηκαν ότι καλό θα ήταν ίσως να έχουμε ε, κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο που είναι διαλειτουργικό. Κάτι που δεν το έχουμε ακόμη βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Εγώ σας ερωτώ μετά από όλα αυτά, πέραν των μεγάλων και ευσεβών πόθων, πραγματικά τι μπορούμε να περιμένουμε τα επόμενα τρία χρόνια για να μπορεί να είναι πραγματικά επιχρησιακός ο οργανισμός και να μην παράγει απλά γραπτά και συστάσεις, πολύ καλε όλες βέβαια, αλλά εντελώς ε, θεωρητικά, ε, σε θεωρητικό επίπεδο, μη λειτουργικέ, μη επιχειρησιακέ. Okay. In absence of... άλλων ερωτήσεων, να κάνω και εγώ τη δική μου. Πρέπει να σας πω ότι διαρωτώμε. με λέγω. Υπάρχει πλήρης αντίληψης του ζητήματος της ενίας του ΠΕΣΚΟ αυτή η συνεργασία στην άμυνα μεταξύ κρατών μελών. Όταν το συζητούμε μου δημιουργούνται βασικά ερωτήματα αν υπάρχει κοινή αντίληψη των απειλών. Ο κ. Νάτς που μίλησε προλίγου αναφέρθηκε στο ότι δεν πιστεύει στη ρωσική απειλή. Και αυτό αποδεικνύει, αποδεικνύει αυτό που θέλω να πω και τις ανησυχίες μου. Διότι βέβαια συμμερίζομαι την άποψη του κ. Νάρτς για τους φοβερούς κινδύνους εκ Μέσης Ανατολής και εκνότου. Αλλά σίγουρα υπάρχει και πρόβλημα και κίνδυνος από Ανατολάς. Και πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Να ληφθεί εξίσου υπόψη. Κύριε Ντόμεκ, είπατε ότι οι υπουργοί θα πρέπει να εξετάσουν τη μακροπρόθεσμη αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Την άνοιξη θα γίνει αυτό του 2019. Πολύ απέχει αυτή η ημερομηνία. Εν τω μεταξύ υπάρχουν διάφορες μορφές συζητήσεων και πολλά προγράμματα που προωθούνται. Τώρα διαρωτώ με μήπως θα πρέπει αυτή η συνάντηση να γίνει πιο πριν, να γίνει αυτή η αξιολόγηση νωρίτερα, να εξεταστούν οι εξελίξεις. Ελπίζω, ελπίζω έτσι να γίνει. να γίνει μια επίσημη πλήρης διεξοδική ανάλυση. Να ληφθούν αποφάσεις. Ποιο είναι το ακριβές περιεχόμενο των προγραμμάτων που θα αναπτυχθούν με τη Σερβία. Εγώ ανησυχώ πολύ για το θέμα της ασφαλείας των Βαλκανίων. Όλοι μας πιστεύω ανησυχούμε γι' αυτό. Θέλουμε να καταβάλουμε προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα. Πιστεύουμε ότι είναι άκρος αναγκαίο. Αλλά πρέπει να πω ότι θυμόμαστε ακόμα το πεδίο που προσπαθούμε να καλύψουμε. Το πεδίο και το βάθος συνεργασίας Σερβίας με χώρες όπως είναι η Ρωσία. Το τονίζουμε αυτό σε εκθέσεις μας. Όπως την πρόσφατη έκθεση Μακάλιστερ περί Σερβίας. Αναφέρουμε τις ανησυχίες μας για τις σχέσεις Σερβίας-Ρωσίας. Κυρίως στη στατιστική, στατιωτική συνεργασία με Λευκορωσία, Ρωσία, συμμετοχή σε κοινέ ασκήσεις στατιωτικές και θέλω να ξέρω ποιες είναι οι απόψεις σας όσον αφορά το βαθμό συνεργασίας στον αμυντικό τομέα με τη Σερβία. Ευχαριστώ. Κύριε Ντόμακ, απαντήστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλα τα μέλη. Και για τις ενθαρρύνσεις και για τις ερωτήσεις. Το θέμα της συνεργασίας στο ΠΕΣΚΟ που έθεσε εκεί η Πρόεδρος και ο κύριος Γκάλερ Ποια είναι η βασική αντίληψη. Η αμυντική συνεργασία είναι ένα εργαλείο. Θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερη ε, συνοχή στον αμυντικό συνδυασμό των κρατών μελών. Τι εννοώ. Υπάρχει κατάλογος κριτηρίων και υποχρεώσεων, επί των οποίων πρέπει να συμφωνήσουν. Αυτός ο κατάλογος πρέπει να παρέχει υψηλότερο επίπεδο αμοιβαίων δεσμεύσεων μεταξύ των κρατών μελών που επιθυμούν να συμμετάσχουν. Επανειλημμένα είπα ότι τα προγράμματα που θα απορρεύσουν από το ΠΕΣΚΟ δεν είναι το σημαντικότερο τμήμα της συνεργασίας. Οι δεσμεύσεις των κρατών μελών για να μπουν σε αυτό το ομόρφωμα μεσοπρόθεσμα οδηγεί σε μια ολοκλήρωση αμυντική. Αυτό θα δώσει συνοχή πολιτική, επιχειρησιακή και βιομηχανική. Όπως γνωρίζετε, σε αυτό το στάδιο διεξήχθησαν συζητήσεις με τα κράτη-μέλη όσον αφορά τα κριτήρια. Είχαμε οργανώσει εργαστήρια. Τον επόμενο μήνα, αρχές του επόμενου μήνα, θα συζητήσουμε τη διακυβέρνηση και τη δίκηση. Και αργότερα, Οκτώβριο, τα διάφορα προγράμματα που έχουν προωθηθεί, έχουν υποπληθεί από τα κράτη-μέλη. Έχουμε περίπου 36, ίσως να έρθουν κι άλλα. Όπως λέω όμως, πρέπει τώρα να συγκεντρωθούμε περισσότερο με τη διακυβέρνηση του συστήματος, με τα κριτήρια. Περισσότερο από τα προγράμματα που είναι απόρρια του ΠΕΣΚΟ. Και πιθανότατα καταθάσουν και άλλα προγράμματα στο μέλλον. Αν δούμε το χρονοδιάγραμμα που μας έδωσε το Συμβούλιο τέλος του έτους, αρχές επομένου έτους, θα έχουμε απόφαση του Συμβουλίου για την ΠΕΣΚΟ. Στο μέλλον, το ΚΑΡΤ θα βοηθήσει να εντοπίσουμε άλλα προγράμματα, τα οποία αξίζουν να υλοποιηθούν στα πλαίσια του περιβάλλοντος ΠΕΣΚΟ. Αυτά λοιπόν για το ΠΕΣΚΟ. Τώρα, μια άλλη ιδέα που επανειλημμένα αναφέρεται σε εκθέσει και πιο πρόσφατα στην έκθεση του Μαρτίου. Δηλαδή, ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα χρηματοδοτείται τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Αυτό συζητήθηκε στη μακροπρόθεσμη αναθεώρηση με του ε, υπουργού και του ΕΡΠΑ. Υπήρξε ενδιαφέρον να προωθηθεί η ιδέα στο βαθμό που δεν υπονομεύει τη διακυβερνητική φύση του οργανισμού και των αμυντικών ζητημάτων. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση του θέματος. Προχωρώντας την ελοποίηση της μακροπρόθεσμης αναθεωρήσεως και θα είναι σημαντικότατο εν ώψη του επομένου πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου που θα υπάρξει δυνατότητα, αν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το αποφασίσουν, να υπάρξει κάποιο σχετικό κεφάλαιο για διοικητικό κόστος και επιχειρησιακό κόστος του οργανισμού. Σχετικά με το ερώτημά σας, κυρία πρόεδρα δηλαδή, τι θα συμβεί από τούδε και στο εξή μέχρι την άνοιξη του 2019. Γιατί επιλέξαμε την άνοιξη του 2019, διότι το καταστατικό μας, η απόφαση του Συμβουλίου, πρέπει να αναθεωρηθεί το 2019 τώρα και του χρόνου έχουμε αρκετά χαρακτηριστικά που αναδύονται, που είναι σημαντικά, που θα καθορίσουν δεχόμενες αλλαγές όσον αφορά τα καθήκοντα του οργανισμού, όπως την ΠΕΣΚΟ ή το ΚΑΡΔ, παραδείγματα, όπου ο οργανισμός αναλαμβάνει ισχυρότερο ρόλο αμυντικού σχεδιασμού από ό,τι κατά παρελθόν. Υπάρχει και μια λεπτομέρεια, μικρή λεπτομέρεια, το Brexit. και το λαμβάνουμε υπόψη στον καθορισμό του χρονοδιαγράμματος. Πώς θα κινηθούμε στο μέλλον, ποια θα είναι η συνεργασία μας με τρίτα μέρη. Και αυτό είναι σημαντικό. Εν τω μεταξύ, από τούδε και στο εξή, μέχρι αυτή την ημερομηνία θα υπάρξουν συνεδριάσεις με τους υπουργού και τους διάφορους αρμοδίους. Θα τα συζητήσουμε αυτά. Χρειάζεται μεγαλύτερη επαφή μαζί τους και μαζί σας όταν θα γίνει προετοιμασία για την αναθεώρηση Τη αποφάσεως του Συμβουλίου. Είναι μια διαδικασία. Συνεχής. Θα δούμε τι θα του χρόνου. Πώς θα κινηθεί το Διευθύνων Συμβούλιο, το Διευθυντικό Συμβούλιο. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε την ειδική πλειοψηφία και ίσως αυτό να παίξει ρόλο στη λήψη αποφάσεων στον οργανισμό. Για το CARD, όπως είπε και ο κ. Γκάλερ, είμαστε αρχική φάση. Τώρα ξεκινά η διμερής διαβούλευση με τα κράτη-μέλη, ούτω ώστε να λάβουμε τις αναγκαίες πληροφορίες για να προβούμε μετά σε μια ανάλυση, την οποία θα κοινοποιήσουμε σε όλους. Οι πληροφορίες που θα κοινοποιηθούν θα αφορούν, θα, οι πληροφορίε που μα δώσει ένα κράτο μέλο θα αφορά εμά και αυτό το κράτο μέλο. Δεν τα, μέλος, δεν θα τα μοιράσουμε τα στοιχεία αυτά στα άλλα κράτη-μέλη. δεν ήταν αρκετά ανοιχτά τα κράτη-μέλη μέχρι τώρα, δεν έδιναν όλε τι αναγκαίε πληροφορίε. Αυτή ήταν η πρώτη εντύπωσή μου. Πρώτη εντύπωση. Επέμεινα. Ότι χρειάζονται διάφορα στοιχεία. Όχι μόνο οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου. Θα πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας από πλευρά 22 κρατών μελών που είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, αυτά τα κράτη-μέλη να Μα λένε πώ κινούνται στον αφορά τον αμυντικό σχεδιασμό του ΝΑΤΟ στα πλαίσια τη κοινή διαβούλευση ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Όταν θέλουμε να έχουμε συνοχή, να υπάρχει συντονισμό μεταξύ του τι κάνουμε εδώ και εκεί, όλα εξαρτώνται από το επίπεδο διαφάνεια ε, που θέλουν να υλοποιήσουν τα κράτη-μέλη. για το οποίο και θα επανέλθω αργότερα με του συναδέλφου τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο επόμενο σημείο. Ένα σημαντικό στοιχείο ο κ. Πάσκου θα το έθεσε. Το θέμα του κόστου. Συμφωνώ. Όλα αυτά τα εργαλεία θα λειτουργήσουν μόνο αν υπάρχει εμπιστοσύνη, μάλλον όχι κόστο, ζητά συγγνώμη διερμηνέα. Εμπιστοσύνη. Και τα χρήματα δεν θα αλλάξουν την κατάσταση. Η εμπιστοσύνη μεταξύ κρατών μελών παίζει ρόλο. Και οι δεσμεύσει που θα αναλάβουν σε υψηλό επίπεδο μέσω τη ΠΕΣΚΟ, εκεί θα γίνει διαφορά. όσον αφορά αυτά που είπε ο κ. Τι περιμένω στην πραγματικότητα. Ελπίζω ότι προχωρώντας δεν λέω ότι αυτά που κάναμε ήταν απλά ρητορικά σχήματα και λόγια. Θα ήταν άδικο κάτι τέτοιο. Έναν των προκατόχων. Αλλά υπολείπεται των δυνατοτήτων του οργανισμού. Τι λέει η συνθήκη αμυντικές δυνατότητες, έρευνα, κοινή, κοινός εφοδιασμός, εξοπλισμός. Περίπου 40% των αναμενωμένων κάναμε για τα δύο πρώτα στοιχεία, ελάχιστα στο τρίτο στοιχείο και σχεδόν τίποτα στο τελευταίο κομμάτι. Αν θέλουμε να κινηθούμε σωστά, αυτό εξαρτάται από το πόσο θα εφαρμοστούν και άλλες δραστηριότητε. Τι βλέπω ότι είναι σημαντικό τώρα να έχουμε χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ενώσεω. Αυτό δεν αρκεί όμως για να κινηθούμε σωστά και σε σωστή κατεύθυνση. Σε ύψιστο επίπεδο υπάρχει πρόθεση από του αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων. Θέλουν η ευρωπαϊκή διάσταση να προωθείται σφαιρικά, σε παγκόσμιο επίπεδο. Και δεν έχουμε πολύ χρόνο να καλύψουμε τα ελλείμματα τη βιομηχανική βάση Πρέπει να εγκαταλειφθούμε την ευκαιρία τώρα για να το πετύχουμε αυτό. Τι ελπίζω. Ελπίζω ότι το ΠΕΣΚΟ θα κάνει την αλλαγή για την αμυντική οργάνωση της Ευρώπης. Και το CARD θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στα σοβαρά. Κάτω παρελθόν, όταν θέλαμε να σχεδιάσουμε την ανάπτυξη δυναμικότητας, δεν λέω ότι τα, τα, κάναμε στραβά, αλλά τα κράτη-μέλη δεν έλαβαν υπόψη την πτυχή στο δικό τους εθνικό μυντικό σχεδιασμό. Αν πάω στην περίοδο που ήμουν στο ΝΑΤΟ, η διαδικασία μετικού σχεδιασμού του ΝΑΤΟ κράτης είχε αρχίσει πολύ πιο παλιά. Αλλά λάβετε υπόψη ότι χρειάζεται συμμετοχή μεγαλύτερη των κρατών μελών για να πετύχουμε τους στόχους. Πολιτικός πώς υπάρχει η βούληση πρόοδου. Τέλος η σχέση με τη Σερβική Δημοκρατία. Υπογράψαμε συμφωνία συνεργασίας. Διοικητική διευθέτηση το 2012. Όπως προανέφερα, αν έχουμε αυτές τις διευθετήσεις, δεν πρέπει να είναι μόνο λόγια. Πρέπει να πετυχαίνουμε το σκοπό μας. Ανάπτυξη δυνατοτήτων των κρατών μελών, που θα είναι κάτι εποφελές και για, τα, και για το άλλο μέλος που συμβάλλει στην ΚΕΠΑ. Η Δημοκρατία της Σερβίας θα συμβάλλει στην ΚΕΠΑ, αλλά για κάθε συγκεκριμένη δραστηριότητα και χρειάστηκε κάποιος χρόνος ούτω ώστε η Δημοκρατία της Σερβίας ενεργά να συμμετάσχει στις ομάδες αμυντικές, στις μονάδες αμυντικές, όταν έφτασα το 2015 στη θέση αυτή, η Δημοκρατία της Σερβίας δεν συμμετείχε σε καμία δραστηριότητα. Απλώς ένα κενό, ένα χαρτί ήταν η συμφωνία. Θα συμμετάσχουν κατά περίπτωση όταν τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι η συμμετοχή της Σερβίας δίνει προστιθέμενη αξία. Είναι θέμα πρακτικό περισσότερο. Εξετάζεται η δυνατότητα, Φερρυπίν, σε προγράμματα που αφορούν την καταπολέμηση αυτοσχεδίων εκρηκτικών μηχανισμών, που είναι κάτι πολύ σημαντικό στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, να υπάρξει συνεργασία. Εκεί δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος να ακολουθηθεί λάθος κατεύθυνση. Η διοικητική διευθέτηση, όπως είπα επανειλημμένα, είναι απλώς μια βάση, μια πλατφόρμα. Και από εκεί θα έχουμε μεγαλύτερη παραγωγικότητα μέσω αυξανόμενης εμπιστοσύνης. Είναι κάτι σαν χρηματιστήριο αν θέλουν τα κράτη-μέλη να αγοράσουν, πρέπει να υπάρξει εμπιστοσύνη. Παράδειγμα, η Νορβηγία, που έχει την παλαιότερη τέτοια συμφωνία. Είναι η έβδομη χώρα όσον αφορά τον αριθμό συνεισφορών και προγραμμάτων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Βλέπετε ότι υπάρχει δυνατότητα, υπάρχουν τα εργαλεία, αλλά πρέπει να αναπτύσσονται και να εφαρμόζονται κατά περίπτωση. Um, uh, με τις παρατηρήσεις αυτής ε, του κυρίου Χόρχερ Ντομέκ θα κλείσω το θέμα αυτό της ημερήσιας διάταξης. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση τα, επί έργων που έχουν σχέση με την άμυνα και τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Και έτσι θα διευρύνουμε τη σύνθεση εδώ του Προεδρείου. Ο, θα υποδεχτούμε τον κύριο Αλέν Αλεξής από τη Γενική Διεύθυνση Πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, το θέμα μας είναι η εφαρμογή της προπαρασκευαστικής ενέργειας για την έρευνα στον τομέα της άμυνας, την οποία ξεκίνησαν τα μέλη της υποπιτροπής μας, της ΣΕΤΕ, και που πλέον έχει εξελιχθεί. Για μία ακόμα φορά ο κύριος Χόρχερ Τόμεκ, ο εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, όπως επίσης και ο κύριος Αλεξής, επικεφαλής της μονάδας που είναι υπεύθυνη για την ε, αεροδιαστημική άμυνα και την αυτιλία της Γενικής Διεύθυνσης GROW της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μαζί μας. Κύριε Τόμεκ και κύριε Αλέξη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε το πιλωτικό πρόγραμμα και η προπαρασκευαστική δράση για την αμυνά ε, ανοίγουν το δρόμο για ένα πλήρες πρόγραμμα ε, ερεύνας στον τομέα της άμυνας. Αυτό το οποίο που μάθαμε από την προηγούμενη προπαρασκευαστική περίοδο είναι πολύ σημαντικά και θα ήθελα να τα αναφέρω εν συντομία. Και θα ολοκληρώσω τη σύντομη παρουσίασή μου με κάποιες παρουσιάσεις επί του πιθανού μέλλοντος της ευρωπαϊκής έρευνας. Ε, θα σας ενημερώσω για το πιλωτικό πρόγραμμα. Το πιλωτικό πρόγραμμα που πρόθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με προπολογισμό 1,4 εκατομμυρίων ευρώ είναι αρκετά προχωρημένο. Ε, όλες οι δραστηριότητες είναι εν εξελίξη αυτή τη στιγμή με ελάχιστες καθυστερήσεις μόνο ενός έως τριών μηνών. Δύο από τις δραστηριότητες θα πρέπει να ολοκληρωθούν στο, στο, στις αρχές του επόμενου έτους το αργότερο, ενώ η επόμενη στο τέλος του 2018. Η προπαρασκευαστική ενέργεια για, τον τομέα της, για την έρευνα στον τομέα της άμυνας είναι μια πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια, έχει μεγαλύτερο προπολογισμό, ε, ε, έχει τρία προγράμματα εργασίας, αλλά οι δραστηριότητες θα διαρκέσουν περισσότερο. Ο εγκεκριμένο ε, προπολογισμό του 2017 είναι 27 εκατομμύρια, το 2018 έχουν ζητηθεί 40 εκατομμύρια και πάλι 25 εκατομμύρια το 2019. Το συνολικό ποσό των 90 εκατομμυρίων ευρώ θα μας επιτρέψει να δοκιμάσουμε διάφορα εργαλεία, τομείς και χώρους έρευνας και να βελτιώσουμε ως εκ τούτου την κατανόηση που έχουμε για το ποιο θα πρέπει να είναι στο μέλλον ένα παραγωγικό πρόγραμμα ε, άμυνας ε, της ε, Ευρώπης. Έτσι δεν, αν περιοριστούν οι πόροι δεν θα μπορέσουμε να διερευνήσουμε ε, όλους τους τομείς και αυτό θα ε, φανεί στο αποτέλεσμα. Ε, τρέχον πρόγραμμα, την προπαρασκευαστική, η προπαρασκευαστική δράση χρηματοδοτεί τρεις τομείς. Την τεχνολογία για ε, ε, ενισχυμένη επιχειρησιακή γνώση, προγράμματα πέρα από τα υφιστάμενα και τον προγραμματισμό. Ε, η, τελική προθεσμία υποβολής προτάσεων θα λήξει στο τέλος της εβδομάδας ενώ για το ε, θέμα της τεχνολογικής επίδειξης θα ολοκληρωθεί στο τέλος Οκτωβρίου. Με αυτόν τον τρόπο έχει στηθεί μια επιτροπή αξιολόγησης με μέλη από άλλους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά πάσα πιθανότητα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίοι θα σταθμίσουν και θα αξιολογήσουν τις προτάσεις με τη βοήθεια ε, ε, ανεξάρτητων ειδικών. Στο τέλος του χρόνου ή στη χειρότερη περίπτωση τον Ιανουάριο του 2018 σκοπεύουμε να υπογράψουμε την βασική συμφωνία και μετά τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου θα δημοσιεύσουμε και τις νέες προσκλήσεις ενδιαφέροντος που κατά πάσα πιθανότητα θα δημοσιευθούν το πρώτο τρίμηνο του 2018. Το ίδιο χρονοδιάγραμμα αναμένεται και για την τρίτη και τελευταία ομάδα προσκλήσεων που αναμένεται να ε, δημοσιευθεί το πρώτο τρίμηνο του 2019. Εν γέννη, με έχω την χαρά να αναφέρω ότι έχουμε ε, ε, ε αυτά όλα αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα είναι ενθαρρυντικά. Και τώρα θα ήθελα να πω δύο λόγια για τα όσα αποκομίσαμε. Ε, έχουμε παραγωγική βοήθεια με την ε, θέση προτεραιοτήτων των προτάσεων Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη σύνταξη τεχνικών ε, περιγραφών και ως εκ τούτου ο οργανισμός μας είναι το επίκεντρο ε, της προσπάθειας αυτής όπως έχει ζητηθεί από τους υπουργού Άμυνα το Μάιο. Αυτή τη στιγμή οι δομές μας έχουν δείξει ότι είναι απολύτως κατάλληλες για να χειριστούν τα θέματα αυτά. Η πρακτική εφαρμογή γίνεται και στο πιλωτικό πρόγραμμα και στην προπαρασκευαστική ε, ενέργεια. Ε, το περασμένο Σεπτέμβριο έχουμε δημιουργήσει μία μονάδα ε, προπαρασκευαστικής ενέργειας που από τον Ιανουάριο θα αποτελείται από πέντε μέλη. Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι για πρώτη φορά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας διαχειρίστηκε χορηγίες και για πρώτη φορά χρησιμοποιήσαμε ε, ε, εργασία πληροφορικής και έρευνας. Έτσι λοιπόν ο Ευρωπαϊκός ε, Οργανισμός Άμυνας ε, παίζει έναν σημαντικό ρόλο τόσο ε, ανάντι όσο και στην υλοποίηση. Δεύτερη παρατήρηση και για την προπαρασκευαστική ενέργεια και για το μελλοντικέ δράσει του προγράμματος οι ρόλοι των διαφόρων παραγόντων που θα συμμετάσχουν θα πρέπει να ξεκαθαριστούν σαφώς. Η επιτροπολογία, παραδείγματο χάρη, θα ε, ε, ε, ισχύσει και θα εμπλακεί η Επιτροπή και η αρμόδια Επιτροπή του προγράμματος. Αλλά πρέπει να υπάρξει η υλοποίηση ενός ρόλου για τον οργανισμό. Θα πρέπει όμως ο ρόλος αυτός να είναι παραγωγικός και να ληφθεί και να φροντίσουμε να υπάρχει ένα πρόγραμμα ε, που θα δώσει σωστές προτεραιότητες στον τομέα, στους τομείς της έρευνας και θα εξασφαλίσει τις διάφορες προτεραιότητες που έχουν συμφωνήσει τα κράτη-μέλη στην ανάπτυξη δυνατοτήτων. Ταυτόχρονα θα πρέπει αυτό να συνάδει με τις αμυντικές ανάγκες του ε, ΝΑΤΟ. Θα πρέπει να ε, ληφθούν αποφάσεις βέβαια σε θέματα επιλογής. Θα είναι λοιπόν απολύτως λογικό να αναγνωριστεί ο σημαντικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας έτσι ώστε να γίνει σωστή κατανομή των ρόλων και να συνεισφέρουμε στην επιτυχία του εγχειρήματο. Και αυτό είναι ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να υπογραμμίσω ο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Άμυνας θα δικαιολογείται πολιτικά αν αναπτυχθεί και φανεί παραγωγικό ε, και δώσει πραγματικ... Ε, προγράμματα πραγματικών δυνατοτήτων που θα χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας και το Ευρωπαϊκό ε, Ταμείο Άμυνας συνολικά δεν θα πρέπει να είναι ούτε να θεωρούνται ότι είναι επιδότηση προς τη βιομηχανία. Το Ταμείο θα πρέπει να δώσει δυνατότητες που θα έχουν προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη και που δεν θα μπορούσαν να προχωρήσουν τα κράτη-μέλη μόνο τους και θα πρέπει να διευκολύνουν τους πολίτες. Και γι' αυτό είναι σημαντικό ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας να συνεισφέρει την προσπάθεια αυτή με χρήση της εμπειρίας, της τεχνογνωσίας και όλα όσα συζητήσαμε στην προηγούμενη συνεδρία. Η γενική, ε, η γενική στρατηγική της, της, ε, ε, της έρευνας στον τομέα της άμυνας, παραδείγματος χάρη αυτή τη στιγμή κάποια από αυτά τα στοιχεία λείπουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ταυτόχρονα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας είναι βασικός υποψήφιος για την υλοποίηση και μπορεί να προσφέρει την εμπειρία του πιλωτικού προγράμματος των, ε, των ε, ενεργειών ε, ε, ε, των παραπροσκευαστικών ενεργειών. Και ίσως είναι κατάλληλη στιγμή να πούμε ότι η συνολική αξία της, των έργων τεχνολογίας, ε, τεχνολογίας και έρευνας είναι περίπου ένα δις ευρώ. Και όπως είπα και πριν, αυτή τη στιγμή υποστηρίζουμε περίπου 100 προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας. Και τέλος, για να μπορέ... είμαστε σε θέση να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή χρήση αυτών των προγραμμάτων, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Η πρόσληψη, η αποδοχή από τα κράτη-μέλη των αποτελεσμάτων της έρευνας θα είναι το τελικό μέτρο της αξίας της. Είτε γίνει μέσω άλλων προγραμμάτων, είτε μέσω ε, εθνικών προγραμμάτων και έργων, η αποδοχή είναι απαραίτητη για να συνεχίσει η έρευνα σε μελλοντικές δυνατότητες. Θα κλείσω την παρουσίασή μου λέγοντας ότι ε, το πιλωτικό πρόγραμμα και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες αποτελούν χρήσιμες ε, ενέργειες εν ώψη της συνέχισης της Ευρωπαϊκής Έρευνας στον τομέα της άμυνας. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας έχει την δυνατότητα να παίξει έναν σημαντικό ρόλο ανάντι ε, στον χώρο της έρευνας και αυτό πρέπει να αναγνωριστεί εκτεταμένα. Και αυτό σημαίνει, επαναλαμβάνω, ότι ο κλάδος είναι ε, κατάλληλος για να συνεισφέρει στο πρώτο αυτό πρόγραμμα έρευνας. ΣΕΚ. Πρέπει να το κάνει αυτό. Και επαναλαμβάνω την μακροπρόθεσμη αναθεώρηση που ενέκραν οι Υπουργοί, ότι ε, η υλοποίηση, ε, θα επέλθει έτσι η υλοποίηση του μέλλοντος που όλοι βλέπουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης δεν υπάρχει ανάγκη δημιουργία νέων δομών για να γίνουν εργασίες όπως οι ανάντι ε, εργασίες. Αναφέρουμε παραδείγματο χάρη στην πρόταση της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας στην Άμυνα που θα επαναλάβει απλώς αυτά που γίνονται από το 2004. Θα, ήταν πιο λογικό και από την άποψη οικονομίας και αποτελεσματικότητας να χρησιμοποιηθούν οι δυνατότητες του οργανισμού. Και συγκεκριμένα έχει αναφερθεί αυτό σε διάφορες εκθέσεις. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Ντόμεκ και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Αλέα Αλεξής από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΓΚΡΟ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω την κατάσταση ό,τι αφορά την εφαρμογή του πιλωτικού σχεδίου και των προπληκτικών σχεδίων και των παραπαρασκευαστικών ενεργειών εν αγωγή, κάτι μπορεί από πολλε πλευρές να είναι ενδιαφέρον, θα ήταν να βάλουμε στην, στο πλαίσιο αυτών των δράσεων στον τομέα της άμυνα. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα defense action plan, ε, ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, με στόχο να μην δοθεί σημασία μόνο στην ανάπτυξη, στην άμυνα, αλλά στην αλυσίδα συνολικά. Γιατί ο στόχος, οπότε το στόχος, δεν είναι η έρευνα αυτή καθεαυτή, αλλά οι δυνατότητες. Γι' αυτό λοιπόν την αλυσίδα, τη γενική αλυσίδα, τη βλέπουμε ολιστικά. Δηλαδή χρηματοδότηση της έρευνας, μια πτυχή δεύτερο. Ανάπτυξη και δυνατότητες και βλέπουμε και κάποιες επιλογές για την ανάπτυξη γενικών δυνατοτήτων. Γιατί αλλιώ χάνουμε το στόχο, τον πολιτικό στόχο που είναι η ανάπτυξη δυνατοτήτων. Επί της ουσίας, προτείνουμε δύο windows, window research και window capacity. Αυτά τα δύο παράφερα. Και στο δεύτερο, τον Ιουνίο, κάναμε μια πρόταση κανονισμού για την ανάπτυξη που μελετάται στη στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συγγνώμη, και το Συμβούλιο. Δεν θα αναφέρω κάτι παραπάνω και έρχομαι στο κομμάτι της ε, έρευνας όπου έχουμε τα πιλωτικά προγράμματα και θα έχουμε και τα πιλωτικά προγράμματα του 2021. Για τα πιλωτικά προγράμματα, πρώτα απ' όλα. Το πιλωτικό πρόγραμμα. Ήδη αναφέρθηκαν τα τρία ζητήματα, τα τρία θέματα, παρά τον προπολογισμό που είναι σχετικά περιορισμένος κάτω από 1,5 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή, έχουμε ε, παρόλα αυτά μεγάλη επιτυχία σε επιχειρήσεις, γιατί έχουμε πάρει 21 προτάσεις. Άρα ενδιαφέρον υπάρχει από την ε, βιομηχανία. Επίσης έχουμε λάβει προτάσεις ποιοτικέ, κάτι που δείχνει το ενδιαφέρον του τομέα. Και κάτι άλλο σημαντικό είναι ότι κοινοπραξίες εκπροσωπούν 8 διαφορετικές χώρες. Υπάρχει λοιπόν ευρωπαϊκή διάσταση. Ξεκάθαρα. Δεν έχουμε μια-δυο επιχειρήσεις από ένα ή δύο κράτη-μέλη, αλλά μια δυο ή δύο κρατή μέλη, αλλά απο προσέγγιση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Επίσης σημαντική είναι και η συμμετοχή των ΜΜΕ και ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, τα οποία εκτέλεσαν ενδιαφέρον. Κάτι επίσης πολύ ενθαρρυντικό για το μέλλον. σε ό,τι αφορά την προπαρασκευαστική ενέργεια, που είναι και το βασικό θέμα. Ξεκίνησαν οι εργασίες, θα έρθουν, θα έρθουν σιγά σιγά προτάσεις, έχουν ξεκινήσει δηλαδή οι διαγωνισμοί, έχουμε ε, το demonstrator για τα ναυτικά, το δεύτερο είναι η προστασία για τα συστήματα των στρατιωτών, ένα θέμα είναι η τεχνολογική πτυχή για το μέλλον, ένα εκατομμύριο πολύ σημαντικά τα θέματα αυτά, γιατί μπορούμε να έχουμε πολλές επιχειρήσεις και κοινοπράξεις που θα συμμετέχουν σε αυτή την παρασκευαστική ενέργεια που δεν γίνεται μόνο για λίγες επιχειρήσεις ή για λίγα κράτη-μέλη. Αντίθετα δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σε ένα μεγάλο φάσμα επιχειρήσεων για τους κανόνες συμμετοχής, όπως ξέρετε, αναθεωρήθηκαν για να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες του τομέα της άμυνας. Ακόμη και στο μη στρατιωτικό τομέα πρέπει να ληφθούν υπόψη ιδιαιτερότητες για τις συμμετοχές. Έχουμε ζητήσει πέντε ε, φορείς από πέντε διαφορετικές χώρες για να έχουμε ευρωπαϊκή διάσταση. Και στα υπόλοιπα τρεις φορείς ε, που θα εκπροσωπούν διαφορετικά κράτη. Θέλουμε όμως αυτή τη διασυνοριακή διάσταση, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό. Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις που μπορούν να συμμετέχουν. Πρόκειται βέβαια για επιχειρήσεις κρατών μελών, να εξαίρεση την Νορβηγία. Έχουμε τη δική συμφωνία με τη χώρα αυτή. Με τη χρηματοδοτική συμμετοχή της Νορβηγίας βέβαια, αν θέλει να συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα. Οι ειδικοί κανόνες συμφωνήθηκαν σε ό,τι αφορά τη μη διάδοση των αποτελεσμάτων στον μη στρατιωτικό τομέα. Διάδοση αποτελεσμάτων, αλλά στον αμυντικό όχι. Υπάρχει επίσης απαγόρευση μεταφοράς των αποτελεσμάτων ε, κοινοποίησης τους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε λοιπόν να διατηρήσουμε όλα αυτά τα αποτελέσματα στο ευρωπαϊκό πεδίο. Και επίσης ε, για το EPR έχουμε στου κανόνες. Ε, το συζητήσαμε με τα κράτη-μέλη το λεπτό αυτό θέμα και με τις επιχειρήσεις. Συμμετέχοντες παραμένουν λοιπόν ε, κάτοχοι των δικαιωμάτων πραγματική διοκτησίας. Η Ένωση βέβαια έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στα αποτελέσματα στο πλαίσιο του follow-up. Τα κράτη-μέλη επίσης μπορούν να λάβουν μια ειδική έκθεση για τα IPR τα πιο εμπιστευτικά στοιχεία δεν θα τα περιλαμβάνουν, αλλά θα μπορούσαν να ενημερωθούν τα κράτη-μέλη παρόλα αυτά. Και σε περίπτωση follow-up, αν αποφασιστεί κάτι τέτοιο από κρατημέλη, κράτη-μέλη, λοιπόν, αυτά τα κρατημέλη θα μπορούν ε, δωρεάν να επωφεληθούν το IPR για την άνοιξη του προγραμματό του. Τώρα επεξεργαζόμαστε το πρόγραμμα 2018, αύριο πρέπει να ξεκινήσει. Όπως καταλαβαίνετε, από του χρόνου θέλουμε να έχουμε λοιπόν follow-up στο Technological Demonstrator, αυτό είναι το βασικό πρόγραμμα, για να μπορέσει να καταλήξει. 40 εκατομμύρια προπολογισμό πρέπει να εξασφαλιστεί αυτό το ποσό για να μπορέσει να συνεχιστεί η εργασία. Ποια είναι τα πρώτα διδάγματα που αντλούμε. Σύντομη είναι η χρονική περίοδος, μόνο κάποιοι μήνες. Κάποια πρώτα Διδάγματα όμως έχουμε αντλήσει. Σε ό,τι αφορά τα θέματα που επελέγησαν για την προσκευαστική ενέργεια. Δείχνουν μεγάλη πραγματική προσθέμενη αξία στην έρευνα σε αμυντικά θέματα. Δεν είναι έρευνα για πρώτα δι της χρήσης, αλλά για αμυγός αμυντικά προϊόντα. Βλέπουμε μεγάλη συμμετοχή των κρατών μελών στο πλαίσιο της επιτροπολογίας. Πάρα πολύ ενεργά τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την ε, προετοιμασία του προγράμματος εργασίας. Και ο οργανισμός άμυνας έχει σημαντικό ρόλο. Αλλά και η διαδικασία επιτροπολογίας είναι σημαντική και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει και αυτό το λόγο του και θα συμμετέχει πλήρως στη διαδικασία. Σε ό,τι αφορά τις όρους διακυβέρνησης, έχουν προσαρμοστεί στο ειδικό αυτό τομέα της άμυνας με την επιφύλαξη ενδεχόμενων βελτιώσεων, τροποποιήσεων για το πρόγραμμα του 2018. Δηλαδή δεν έχουμε ακόμη αποκτήσει επαρκή απόσταση για να μπορούμε να κρίνουμε. Ε, βλέπουμε καλή συμμετοχή ε, των επιχειρήσεων, δείχνει η συμμετοχή τους ότι ενδιαφέρονται Μιλάμε για τις επιχείρησεις που συμμετέχουν στις κοινοπραξίες. Υπάρχει λοιπόν ενδιαφέρον επιχειρηματικό. Θεωρούμε ότι σε αυτή τη φάση η προπαρασκευαστική ενέργεια και το πλωτικό πρόγραμμα είναι επιτυχή, με την επιφύλαξη βέβαια των μελλοντικών εξελίξεων και το τι διδάγματα θα μπορούσαμε να αντλήσουμε. Ε, αυτό θα είναι πολύ σημαντικό ενώ το 2021. Είναι λίγο πρόωρο τώρα να καταλήξουμε σε τελικά συμπεράσματα. Αυτά είναι ο λίγης ε, πώς έχει κατάσταση, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα ευχαριστήσω και τους δύο δικαιοκριμένους ομιλητές του πάνελ. Θα ξεκινήσουν οι ερωταπαντήσεις και ο κύριος Γκάλερ ξεκινάει πρώτος. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, περιμένω. Θα ήθελα σε σχέση με το τελευταίο να κάνω μια ερώτηση. Έχουμε αυτά τα διάφορα στάδια, πιλωτικό πρόγραμμα ε, και σίγουρα υπάρχει μια λογική ακολουθία. Το ερώτημά μου τώρα είναι αν μπορούμε ήδη από τώρα για την προπαρασκευαστική ενέργεια να έχουμε κάποια διδάγματα που έχουν αντληθεί από το πιλωτικό πρόγραμμα. Ήδη δηλαδή αν έχουμε κάποια διδάγματα και σε ό,τι αφορά ε, τα μέτρα που θα προετοιμαστούν και θα εφαρμοστούν κατά πόσον έχουμε κάποιες ενδείξεις και κάποιες πληροφορίες για την κατεύθυνση που θα ακολουθηθεί στο βασικό πρόγραμμα. Είχαμε αυτό το Group of Personalities and Defense Research. Είχαμε follow-up. Σε αυτό είναι διαφορετικό ερώτημα. Τι γίνεται σε σχέση με τις συστάσεις αυτής της ομάδας. Και συνολικά, σε ό,τι αφορά αυτά τα διδάγματα Έχουμε και το πρόγραμμα ανάπτυξη ευρωπαϊκή ε, βιομηχανία και θα μπορούσαμε να αντλήσουμε και από εκεί κάποια δάγματα. Έχουμε εμπειρίε. Έχετε κάτι να μα πείτε. Γιατί αν κατάλαβα καλά αυτά που είπατε, ουσιαστικά λέτε ότι είναι πρόωρο ακόμα να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Αλλά κάποια ιδέα η Κομισιόν θα πρέπει να έχει και μαζί με τον Οργανισμό Άμυνα ε, πώ προχωράει το πράγμα και σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και σε συνεργασία με τον ε, Οργανισμό Άμυνας, πιστεύω ότι κάπως έχετε μία ιδέα. Χωρίς να θέλω να προκαταλάβω βέβαια τα πράγματα. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε συνάδελφοι, κάπως διστάζω να σας πρόξω για να ζητήσετε το λόγο. Παρακαλώ σηκώντε το χέρι σας αν θέλετε να μιλήσετε. Ο κύριος Πασκού. Είναι η αρχή. Από την εμπειρία σας μέχρι τώρα. Πόσα προγράμματα κάνουν μια βουλιδοσκόπηση της καταστάσεως. Κατά πόσο αποκρίνονται στις πραγματικές αμυντικές ανάγκες. Μπορείτε να μας πείτε. Μέχρι τώρα βέβαια. Ευχαριστώ. Η κυρία Βαλέρο. Σύντομες ερωτήσεις. Για τα πνευματικά δικαιώματα βρέθηκε λύση. Ήταν πρόβλημα αυτό. Έρευνα μετά. Θα συμπεριλαμβάνονται και τα αυτόνομα απλικά συστήματα τώρα στο εγγύς μέλλον ή στο μακρινό μέλλον. Ευχαριστώ. Δεν ζητά άλλο το λόγο. Θα δώσω το λόγο στα μέλη του πάνελ με την ίδια σειρά που μίλησαν και πριν. Και ίσως να υπάρξει και δεύτερος γύρος ερωταπαντήσεων. Ο κ. Ντόμακ πρώτα. Ευχαριστώ. Για την ομάδα προσωπικότητων θα αφήσω τον κύριο Αλέξη να εξηγήσει. Είναι νωρίς ακόμα για μαθήματα. Κάποια από αυτά τα ανέφερα στην παρέμβασή μου όμως. Το πρώτο. Οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πράγματι δίνουν κίνητρα. Τα κράτη-μέλη και η βιομηχανία έτσι προωθούνται να συνεργαστούν διασυνοριακά. Έτσι πρέπει να χρησιμοποιηθεί το όπλο αυτό. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος εξισώσεως. Το άλλο σκέλος εξισώσεως είναι αυτό που θέσατε κύριε Πάσκου. Παράγουμε αυτά που απαιτούνται. Αυτό είναι το σημαντικό. Πράγματι. Θα το εξασφαλίσουμε αυτό μόνο αν εξακολουθούμε να αναπτύξουμε και την έρευνα και τις δυνατότητες μέσω του σωστού μείγματος διακυβερνητικής μεθόδου και κοινοτικής μεθόδου. Επιτροπολογία δεν αφισβητείται το θέμα η εισρωή στο πρόγραμμα εργασιών ποια θα είναι, βλέποντας τα θέματα που επελέγησαν για τον πρώτο χρόνο. Ανταποκρίνονται στην πρώτη προτεραιότητα που αναφέρεται, στην ενοποιημένη άποψη που υπέβαλαν τα κράτη-μέλη μετά από συζητήσεις στον οργανισμό. Εκμεταλλευόμενοι πλήρω το δίκτυο εμπειρογνωμόνων και τις ομάδες εργασίας που υπάρχουν στον οργανισμό είναι το λογικότερο. Δείχνει σωστό κράμα συζητήσεως για τα κράτη-μέλη και λήψεως σωστών αποφάσεων. Αν δεν κινηθούμε ότι ο τρόπος δεν θα εξασφαλίσουμε ότι το προϊόν των προσπαθειών πραγματικά θα οδηγεί σε αμυντικό εφοδιασμό και προγράμματα δημιουργίας δυνατοτήτων. Μπορεί να έχεις, να έχεις υπέροχα αποτελέσματα που δεν υλοποιούνται, δεν εφαρμόζονται. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογουμένου έτσι και ούτε θέλουμε να υπολοιπόμεθα των στόχων ασφαλείας μας. Σημαντικό τμήμα αυτό. Όσον αφορά τις αμυντικές ιδιαιτερότητες που ανέφερε ο κ. Αλέξης, είναι πολύ σημαντικό. Μπαίνουμε σε έναν τομέα όπου η έρευνα έχει κάποιες αποχρώσεις. Στο μελλοντικό ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα για την άμυνα ίσως πρέπει να εξετάσουμε και πώς διαδίδονται, πώς διαβιβάζονται τα αποτελέσματα, ποια πολιτική θα ακολουθηθεί. Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη αυστηρότητα ενδεχομένω. Άρα κάτι ίσως να αποσαφινιστεί με την πάροδο του χρόνου. Αυτά είναι τα βασικά μαθήματα για σήμερα. Για το ερώτηση κυρία Βαλέρα για την έρευνα. Το αυτόνομο σύστημα ήδη αποτελεί τμήμα του πιλωτικού προγράμματος. Είναι ένα από τα τρία θέματα, τις τρεις δραστηριότητε που προωθούμε. Και στο πρόγραμμα εργασιών του 2018 εμπεριέχεται το πρόγραμμα επίδειξης που αφορά κυρίω τα αυτόνομα αμυντικά συστήματα. Για το IPR θα στραφώ στον κύριο Αλέξη να απαντήσει. Κύριε Αλέξης, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Τα μαθήματα, τα αρχικά. Είναι σύντομη η περίοδος προβληματισμού. να θυμηθούμε το στόχο μας. Δεν θέλουμε να αντικαταστήσουμε τα κράτη-μέλη για την χρηματοδότηση της έρευνας. Η χρηματοδότηση της έρευνας είναι πρωταρχική ευθύνη των κρατών μελών στα θέματα της αμήνης. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία σε κοινοτικό επίπεδο είναι το ερώτημα. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε δύο μαθήματα. Μπορεί να υπάρξει προστιθέμενη αξία όταν συνάδει η δράση με τις προτεραιότητες και δυνατότητες που έχουν καθοριστεί από τα κράτη-μέλη σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή σε περιφερειακό. Πρέπει να συνάδουν με τις προτεραιότητες και δυνατότητες που συμφωνήθηκαν από τα κράτη-μέλη. Καθορισμός προτεραιοτήτων δυνατοτήτων είναι αρμοδιότητα κρατών μελών και όχι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι σημαντικό να υπάρχει συντονισμός μεταξύ αυτών των επιπέδων να λάβουμε υπόψη δε και το ΠΕΣΚΟ. Γι' αυτό στο πρόγραμμα ανάπτυξης που προτείναμε, ε, προτείνουμε και ένα μπόνους. Θα δείτε στα πλαίσια του ΠΕΣΚΟ. Και πρέπει να γίνεται διαφοροποίηση ε, όσον αφορά τη συνεργασία. Δεν είναι τόσο εύκολη σε αμυντικά ζητήματα, συνεργασία. Ένα από τα μέσα ε, να ευνοήσουμε τη συνεργασία είναι η υποστήριξή της, οικονομικός. Τα είδαμε στα πιλωτικά προγράμματα και στην προπαρασκευαστική δράση το είδαμε να ισχύει. Τρίτον, δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό παρά μόνο αν συμμετέχουν όλοι. Τι σημαίνει, κράτη-μέλη, βιομηχανία και να υπάρχει στενή διασύνδεση μεταξύ των δύο για τα κοινοτικά προγράμματα επιμένουμε επί του σεβασμού της επιτροπολογίας. Άρα γι' αυτό είμαι πιο επιφυλακτικό από το συνάδελφο όσον αφορά τη κυβερνητική διάσταση. Δεν πρέπει να αναμειγνύουμε την επιτροπολογία και τη διακυβερνητική πτυχή. Όμως, ο ρόλος των κρατών μελών είναι θεμελιώδου σημασία. Και στα πλαίσια της επιτροπολογίας για την προετοιμασία των προγραμμάτων εργασίας διότι τα κράτη-μέλη δίνουν την τεχνογνωσία τους με την στήριξη των αρμοδίων φορέων. Αλλά είμαστε σε κοινοτικό τομέα και όχι διακυβερνητικό. Τώρα τα προγράμματα που διατηρούνται μέχρι τώρα ανταποκρίνονται πλήρως αυτά στις προτεραιότητες. Γιατί. Διότι συζητήσαμε επί μακρόν με τα κράτη-μέλη στα πλαίσια της Επιτροπής που δημιουργήσαμε, κάθε κάτω μέλος έκανε προτάσεις. Η συζήτηση καμιά φορά ήταν δύσκολη, διότι κάθε κάτω μέλος υπερασπιζόταν φυσικά την πρότασή του, αλλά επέτρεψε αυτή η συζήτηση να διαφανούν προτεραιότητες που ανταποκρίνονται στις ευρωπαϊκές ανάγκες. Για το IPR είναι θέμα δυσχερέστατο. διότι εδώ οι επιχειρήσεις έχουν μια διμερή σχέση με τα Υπουργεία Άμυνας. Και εκεί, σε αυτό το πεδίο, δρούμε διαφορετικά μέσω χορηγιών και επιδοτήσεων. Η ισορροπία που βρέθηκε είναι η εξής. Οι συμμετέχοντες στο consortium για την έρευνα είναι, έχουν την πνευματική διοκτησία. Η Ένωση πρέπει βέβαια να έχει πρόσβαση στα αποτελέσματα για τις ανάγκες μεταγενεστέρων εξελίξεων και αναπτύξεων. Δεν πρέπει να πληρώνουμε δύο φορές το πράγμα. Αν αναπτυχθεί κάτι, πρέπει να έχουμε πρόσβαση στα αποτελέσματα, τα επιτευθέντα. Τα κράτη-μέλη επίσης έχουν πρόσβαση σε μια ειδική έκθεση που συνοψίζει τα βασικά στοιχεία χωρίς να επισέρχεται σε λεπτομέρειες και να αποκαλύπτει εμπιστευτικέ πληροφορίες. Αν εν συνεχεία μια ομάδα κρατών μελών επιθυμεί να συμπεριλάβει αυτό το πρόγραμμα, να το προωθήσει, να το προχωρήσει σε συνεργασία με τη βιομηχανία, αυτή η ομάδα των κρατών μελών θα πρέπει να έχει πρόσβαση δωρεάν σε αυτά τα δικαιώματα διαφορετικά τα κράτη-μέλη και η κοινότητα θα πληρώνει δύο φορές για το ίδιο πράγμα. Κάτι που δεν θα ήταν αποδεκτό. Ευχαριστώ κυρία Αλέξης. Ε, συνάδελφοι, ήταν αρκετά μακροσκελής η παρουσίαση της μακροπρόθεσμης αναθεωρήσεως του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αμήνης και ποια είναι η υλοποίηση της προπαρασκευαστικής δράσεως για την αμυντική έρευνα. Ευχαριστώ τους συγκεκριμένου ε, καλεσμένους μας, μέλη του πάνελ και είμαι σίγουρη ότι και τα δύο θέματα συνεχώς θα συζητούνται από την Υποεπιτροπή μας το επόμενο εξάμεινο και πιθανότατα και αργότερα. Βασιζόμαστε σε εσά να είσαστε παρόντες. Ευχαριστώ πραγματικά πολύ. Θα ξεκινήσουμε σε δύο λεπτά το επόμενο σημείο τη συζήτηση για το επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ, καθίστε. Σας υπενθυμίζω ότι είναι αρκετά βεβαρημένη η σημερινή απογευματινή ημερήσια διάταξη και μερικοί από εμά και για το βράδυ, κατά τη διάρκεια του διευρυμένου Προεδρίου που θα ακολουθήσει. Οπότε ας αρχίσουμε τώρα κατευθείαν. Όπως έχουμε ανακοινώσει κατά την έγκριση της ημερήσιας διάταξης της σημερινής απογευματινής συνεδρίασης, ξεκινάμε σήμερα την προετοιμασία μια σειρά θεμάτων εν ώψη της κοινή μας αποστολής στις Ηνωμένε Πολιτείε και το Norfolk, το ΝΑΤΟ δηλαδή, και ένα από τα σημαντικά ζητήματα που πρέπει να εκτιμηθούν είναι η κατάσταση ασφαλείας στη Μέση Ανατολή. Σήμερα παρουσιάζουμε την, ε, το θέμα από την πλευρά των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Στην προηγούμενη συζήτηση ε, ε, υποσχέθηκα στους συναδέλφους ότι θα μπορέσουμε να προσκαλέσουμε τους εκπροσώπους της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και κάποιους ειδικού των Βρυξελών για να συνεχίσουν την παρουσίαση αυτού του θέματος αργότερα. Πριν όμως πάμε στις Ηνωμένε Πολιτείε, θέλουμε να ε, μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε. Δυστυχώς έγιναν ε, αλλαγές στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και παρά τις προσπάθειες της Γραμματείας δεν καταφέραμε να κάνουμε αυτό που θα θέλαμε να κάνουμε. Θα έχουμε όμως τη δυνατότητα να ακούσουμε εξαιρετικούς ειδικού. Ο πρώτος είναι ο κύριος Ρούλ Μαρκ Γκερέχτ, που είναι κύριος επιστημονικός συνεργάτης του Ιδρύματος για την Πρόσπιση των Δημοκρατιών των Ηνωμένων Πολιτειών και ο δεύτερος ομιλητής θα είναι ο κύριος Γιώση Κούπερ ο οποίος και αυτός είναι κύριος επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου Δημοσίων Υποθέσεων της Ιερουσαλήμ. Προηγουμένως υπήρξε Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Στρατηγικών Υποθέσεων του Ισραήλ. Αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον, καυτό, όπως είπαμε και σε μια από τις προηγούμενες συζητήσεις μας και ως εκ τούτου, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, θα δώσω το λόγο στον ε, κύριο Γκερέχτ πρώτα και στον κύριο ε, Κούπερ Βάσερ μετέπειτα. Oh, <laughs> okay. I, was I was going to let okay. first age wisdom before sorry. <laughs> okay. Λοιπόν, αντιστρέφουμε τη σειρά των ομιλητών. Εγώ έκανα λάθος. Ο κύριος Κούπερ Βάσερ θα πάρει πρώτος το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι τιμή και χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να συζητήσω μαζί σας το πολύ ενδιαφέρον αυτό θέμα. Έχω παρουσιάσει και κάποιες διαφάνειες. Δεν ξέρω από πού προέρχονται, αλλά θα προσπαθήσω να σας τους δείξω, να σας τις δείξω. Θα ήθελα να αρχίσω παραγράφοντας γενικότερα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Τι συμβαίνει, ποιος πολεμάει ποιον. Εν γέννη μπορούμε να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια, Να νάτες οι διαφάνειες, τα τελευταία χρόνια λοιπόν είμαστε ε, μάρτυρες μιας διέρεσης ε, ε, ανάμεσα σε δύο απόψεις στο μουσουλμανικό ε, κόσμο η σχολή των ρεαλιστών και η σχολή των ριζοσπαστών. Οι ρεαλιστές λένε ότι ο μουσουλμανισμός, ο μαμεθανισμός θα πρέπει να ενταχθεί στην ε, υφιστάμενη παγκόσμια τάξη. Ε, ακόμα και αν δεν τους αρέσει θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να ενταχθούν σε αυτήν. Οι ριζοσπάστες ε, πιστεύουν ότι οι μουσουλμάνοι όχι μόνο θα πρέπει να αλλάξουν ταχύτερο δυνατό την παγκόσμια τάξη, αλλά να φροντίσουν να μην επικρατήσουν στην συζήτηση που γίνεται στο μουσουλμανισμό γερμανικό κόσμο οι ρεαλιστές, γιατί ε, στο μυαλό των ριζοσπαστών ο δυτικός πολιτισμός αποτελεί απειλή για το Ισλάμ και δεν μπορεί να γίνει ε, αποδεκτός. Επίσης, ε, γίνεται και πάλι μια διαπάλη στο εσωτερικό του ριζοσπαστικού Ισλάμ μεταξύ δύο διαφορετικών σχολών. Η μία είναι οι υπερ οι οποίοι πιστεύουν ότι η αλλαγή στην παγκόσμια τάξη πρέπει να γίνει άμεσα τώρα, γιατί ήδη η Δύση είναι πολύ αποδυναμωμένη, έχει ε, πέσει σε ειδονισμό και δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έρθει τώρα η αλλαγή. Και τώρα αυτοί που προσπαθούν να φέρουν την αλλαγή το κάνουν μέσω της τρομοκρατίας. Χρησιμοποιούν την τρομοκρατία στη Μέση Ανατολή και στη Δύση για να αλλάξουν την παγκοσμία τάξη τώρα. Υπάρχει τώρα και η άλλη ομάδα, οι ρεαλιστές ε, ριζοσπάστε που λένε ναι, να αλλάξουμε την παγκόσμια τάξη, το χειρότερο δυνατό, αλλά η Δύση, παρότι πραγματικά καθημερινά αποδυναμώνεται, εξακολουθεί να είναι πολύ δυνατή για να τις επιβάλλουμε την αλλαγή στην παγκόσμια τάξη που στηρίζεται στις, ε, ε, στο δυτικό πολιτισμό και στις δυτικές αξίες, να χρησιμοποιήσουμε τη Δύση για να πετύχουμε μια σειρά από ρυθμίσεις που θα μας δώσουν, ε, βοηθήσουν να χρησιμοποιήσουμε τον χρόνο καλύτερα από τον χρησιμοποιεί η Δύση για να, να καταφέρουμε σύντομα να αλλάξουμε την κατάσταση και να αλλάξουμε την παγκόσμια τάξη. Όπως βλέπετε, αν βλέπετε, ποιος είναι σε ποιο στρατόπεδο. Έχουμε και σιίτες και Σουνίτες. Δεν είναι το χάσμα μεταξύ η διαίρεση Σουνιτών Σιητών πιο σημαντική στη Μέση Ανατολή υπάρχει, αλλά η πιο σημαντική διαίρεση είναι ανάμεσα στους, ε, στους πραγματιστές, τους ε, ριζοσπάστες και στους ε, υπερριζοσπάστες. Αυτό είναι ο πραγματικός πόλεμος. Αν το δείτε από τη σκοπιά της δύση, βλέπουμε ότι και στη Δύση υπάρχουν δύο προσεγγίσεις του τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Είναι η ρεαλιστική συντηρητική προσέγγιση, δεν θα μιλήσω για την υπερσυντηρητική, τους τη ρεαλιστική ή συντηρητική θα αναφέρω μόνο, και η φιλελεύθερη προσέγγιση. Και δεν θα μιλήσω για τους υπερφιλελεύθερους, μόνο για τους φιλελεύθερους, γιατί αυτοί έχουν ε, δύναμη. Και τι βλέπουμε όταν ε, εξετάζουμε τη σύγκρουση που εξελίσσεται λόγω των διαφορετικών προσεγγίσεων του τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, είναι το εξή. Ενώ οι ρεαλιστές συντηρητικοί επιδιώκουν καλύτερες σχέσεις με τους πραγματιστές. Οι φιλελεύθεροι είναι εξαιρετικά καχύποπτοι απέναντι στους πραγματιστές και δεν πιστεύουν ότι αξίζει να συνεργαστούν μαζί τους και θα προτιμούσαν να συνεργαστούν με τους ρεαλιστές ριζοσπάστες. Υπάρχει μεγάλη αλλαγή στη Μέση Ανατολή. Η, η, η, οι ηγέτες των ΗΠΑ τώρα έχουν φύγει από τους φιλελεύθερους και προσπαθούν να συνεννοηθούν με τους ε, ε, συντηρητικούς, ε, με τους φιλε... ρεαλιστές ριζοσπάστες. Και είδαμε τι έγινε με το θέμα του Κατάρ και υπάρχει μια μεγάλη διαίρεση σήμερα στη Μέση Ανατολή. Είναι δύο μεγάλες διαφορετικές προσεγγίσεις που κυριαρχούν στη Μέση Ανατολή. Η πιο μεγάλη ε, σημαντική κίνηση της προηγούμενης διοίκησης των ΗΠΑ ε, στην Μέση Ανατολή για να δείξει άνοιγμα και διάθεση συνεργασίας με τους ρεαλιστές ε, ριζοσπάστες ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο πρόεδρος Ομπάμα προώθησε το κοινό ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτό ήταν ένα μεγάλο δώρο που έδωσαν οι φιλελεύθεροι στους Ιρανούς, οι οποίοι υποτίθεται ήταν οι ρεαλιστές ε, ε, ε ριζοσπάστες. Ο Ζαρίφ, ας πούμε, δόθηκε, πήραν αυτό το βραβείο για να δουλέψουν πιο σκληρά έναντι των ε, μουσουλμάνων ριζοσπαστών Όλο αυτό βέβαια δεν ήταν αποτελεσματικό, δεν λειτουργήσε. Αυτή ήταν πάντω η λογική πίσω από τη συμφωνία με το Ιράν. Η συμφωνία με το Ιράν επηρέασε σημαντικά όλη την εικόνα και η αλλαγή της κυβέρνησης των ΗΠΑ διαπιστώνουμε ότι άλλαξε και η προσέγγιση απέναντι στη συμφωνία με το Ιράν και όλα θα εξαρτηθούν από τον τρόπο με τον οποίο ο πρόεδρος Τραμπ θα ε, ε, ανταποκριθεί, θα, έχει, θα ε, αναπτύξει πολιτική σε σχέση με την συμφωνία με το Ιράν. Θα το κάνω και αυτό μέσα στα 15 λεπτά που μου έχουν δοθεί. Θα μιλήσω για αυτήν τη συμφωνία. Γιατί είναι τόσο επικίνδυνη η συμφωνία με το Ιράν. Είναι πολλοί οι λόγοι, οι περισσότεροι από εσά του γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είμαι σίγουρο. Πρώτον, είναι δομημένοι έτσι ώστε ε, έχουν, έχει μια ρήτρα ε, που εξασφαλίζει ότι ε, στο Ιράν ότι έχει ένα νόμιμο τρόπο για τη δημιουργία οπλοστασίου, πυρηνικού οροστασίου. Αυτό είναι το μεγάλο όνειρο των Ιρανών. Στο παρελθόν δεν μπορούσαν οι Ιρανοί να καλύψουν το χάσμα ανάμεσα ε, στο, ε, στον εμπλουτισμό ουρανίου και στην δημιουργία του ε, βόμβας. Τώρα έχουν έναν ασφαλή τρόπο για τη δημιουργία οπλοστασίου μεγάλου, εκατοντάδων ε, όπλων, 20 ή παραπάνω ατομικων βομβών σε πρώτη φάση μέσα, φάση, μέσα σε 15 χρόνια. Τώρα ήδη είναι σε 13 χρόνια. Αυτό ήταν η μεγάλη συμφωνία για το Ιράν. Δεύτερον, έχει πολύ κακή ε, ε, παρακολούθηση, επιτήρηση. Πολύ κακή επιτήρηση. Πράγμα που επιτρέπει στους Ιρανούς ε, να αναπτύξουν στοιχεία του πυρηνικού τους προγράμματος, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζεται να ε, συμμορφώνονται με τη συμφωνία. Κανείς δεν ξέρει τι κάνουν οι επιστήμονες. Δεν υπάρχει παρακολούθηση των Ιρανών επιστημόνων που είναι το πιο ε, σημαντικό στοιχείο, ε, πολύτιμο στοιχείο των Ιρανών. Κάνουν ό,τι θέλουν. Κανείς δεν ξέρει τι κάνουν. Δεν υπάρχει παρακολούθηση του τι κάνουν οι Ιρανοί εκτός του Ιράν. Αν τώρα κάνουν κάτι σε συνεργασία με τη Βόρεια Κορέα ή στη Συρία αυτή τη στιγμή, κανείς δεν το γνωρίζει και κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει. Αυτή η κακή παρακολούθηση άφησαν τους Ιρανούς σε κατάσταση όπου θα μπορούσαν να προχωρήσουν με το πυρηνικό τους πρόγραμμα ακόμα και στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας. Τίποτα δεν γίνεται, δεν συνέβη, ε, κατά της ολόκληρης στρατιωτικής ε, υποδομής, η οποία παρέμεινε άθικτη. Μια εγκατάσταση στο ΚΟΜ, η οποία ήταν περίφημη, γιατί ήταν εξαιρετικά καλά προστατευμένη. Αφέθηκε άθικτη. Όπως και οι άλλες εγκαταστάσεις. Οι φυγόκεντρες που αφαιρέθηκαν από τις εγκαταστάσεις δεν διαλύθηκαν, απλώς φυλάχθηκαν σε κάποια κοντινή εγκατάσταση, σε κάποιο κοντινό χώρο. Όλη η υποδομή εξακολουθεί να υφίσταται και οι Ιρανοί μπορούν να προχωρήσουν ταχύτερα αν αποφασίσουν να εγκαταλείψουν τη συμφωνία. Και μπορούν να το κάνουν από πολύ καλά προστατευμένους χώρους γιατί επιτρέπεται να αγοράσουν ε, σύμφωνα με τη συμφωνία όπλα που θεωρούν απαραίτητα για να αυτοπροστατευτούν απέναντι σε ρωσικά συστήματα ε, ε, μάλλον ρωσικά συστήματα αεράμινας. Επίσης δεν υπάρχει παρακολούθηση των συστημάτων παρακολούθησης. Παράδοσης. Είδαμε τώρα το νέο πύραυλο του Ιράν που εκτοξεύτηκε 2.000 μέτρα. Σε μπορεί να φτάσει και κάποια σημεία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η νέα απειλή του Ιράν που, για την οποία δεν γίνεται τίποτα. Και όλα αυτά τα όπλα, οι πύραυλοι αυτοί αναπτύσσονται για να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές. Δεν πρόκειται να μεταφέρουν ε, απλώς κεφαλές. Δεν υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις στο πρόγραμμα αυτό του Ιράν και στη συμφωνία για το τι θα κάνει το Ιράν επί άλλων θεμάτων, την εξαγωγή της τρομοκρατίας, της, την υποκίνηση ε, εξεγέρσεων σε άλλες χώρες, το να ζητάει την καταστροφή του Ισραήλ κλπ. κλπ. Οι Ιρανοί λοιπόν μπορούν να κινηθούν στην απόκτηση αυτό του οπλοστασίου ε, σε 13 χρόνια χωρίς να αλλάξουν το παραμικρό την πολιτική τους και δεν πρόκειται να την αλλάξουν το τίμημα που θα πάρουμε εμείς από αυτή τη συμφωνία είναι πολύ περιορισμένο. Τα ωφέλη. Ελάχιστα μας δόθηκαν. Ε, παρετήθηκαν από κάποιο από το εμπλουτισμένο ουράνιο που είχαν οι Ιρανοί, αλλά μπορούν να δημιουργήσουν ό,τι θέλουν, ιδίως με τις καινούριες φυγοκέντρους που μπορούν να ε, αναπτύξουν. Μπορούν να παράξουν το, τις ποσότητες που παρέδωσαν ταχύτατα. Κυρίως δε, δεν υπάρχει όριο ε, το, της ποσότητας ε, της πρώτης ύλη που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να παράξουν εμπλουτισμένο ουράνιο. Και τέλος, Σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία, είναι εντελώς αδύναμο να επικρίνει τι κάνει το Ιράν, γιατί πάντοτε φοβάται η Δύση ότι αν κάνει κάτι, οι Ιρανοί θα εγκαταλείψουν τη συμφωνία. Και ως εκ τούτου μπορούν οι, οι, οι Ιρανοί να κάνουν ό,τι θέλουν, να καταλάβουν τη Συρία, την Ιεμένη, να ε, δοκιμάζουν πυράβλους, γιατί η Δύση θα λέει πάντα αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, διότι αν, το, αν κάνουμε κάτι θα ε, ε, ε, καταστραφεί η συμφωνία. Παραδεχόμαστε δηλαδή ότι δεν θέλουμε να φύγουν από τη συμφωνία. Φυσικά, αν δείτε την κατάσταση, θα δείτε ότι το Ιράν θέλει να ε, διατηρήσει αυτή την καταπληκτική συμφωνία που τους δίνει τα πάντα. Σε 13 χρόνια, όταν θα αποκτήσουν αυτό το πλωστάσιο, τότε αυτοί οι ρεαλιστές ριζοσπάστες θα προσπαθήσουν να αλλάξουν την παγκόσμια τάξη στη Μέση Ανατολή, αν δεν ε, το έχουν ολοκληρώσει αυτό μέχρι τότε, και μετά θα προσπαθούν να αλλάξουν την παγκόσμια τάξη του ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό είναι το σχέδιό τους. Και εν το μεταξύ μπορούν να προχωρούν ε, και όλα τους τα υπόλοιπα θέματα χωρίς ε, εμπόδιο. Δηλαδή, το να πούμε ότι το Ιράν συμφωνεί ή μάλλον τηρεί τη συμφωνία είναι ε, παράλογο. Βεβαίως και την τηρεί, διότι δεν καταλαβαίνουν όσοι λένε ότι θα μπορούσαν να μην την τηρεί τι σημαίνει αυτή η συμφωνία για το Ιράν. Το ερώτημα όμως είναι εδώ, τι κάνει για αυτά όλα η Δύση. Το Ισραήλ είναι ένας από αυτούς τους ρεαλιστές συντηρητικούς που ανέφερα στην προηγούμενη μου διαφάνεια. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να απομακρυνθούμε από τέτοιου είδους συμφωνίες με τους ροσπάστες, οι οποίοι το μόνο που θέλουν να επιτύχουν είναι η αλλαγή του, της παγκόσμια τάξη. Εμείς θέλουμε να διατηρηθεί η παγκόσμια τάξη, να διατηρηθεί η σταθερότητα. Και για να το πετύχουμε αυτό είναι να φύγουμε από αυτή τη συμφωνία ή να την αλλάξουμε αν γίνεται. Αν μπορούμε να την αλλάξουμε, καταπληκτικά. Αλλά αν δεν μπορούμε, τότε οι άνθρωποι θα πρέπει να απομακρυνθούν ε, από αυτή την επικίνδυνη συμφωνία, αισθανόμενοι ότι όλα είναι καλά. Ε, αλλά ταυτόχρονα κινούμαστε προς την καταστροφή. Αυτό το είδαμε και στην περίπτωση της Βόρειας Κορέας. Πρέπει να το γνωρίζουμε με ποιο τρόπο θα τα κάνουμε αυτά. Ε, αν πάμε σήμερα στους Ιρανούς, που δεν έχουν ακόμα πυρηνικά όπλα, και τους ζητήσουμε να αναθεωρήσουν τη συμφωνία, θα πούνε όχι, ούτε κατά διάνοια κλπ. Αλλά τελικά θα καταλάβουν ότι δεν έχουν άλλη επιλογή. Όσο πιο ενωμένη είναι η Δύση σχετικά επ' αυτού, τόσο περισσότερα μπορούμε να πετύχουμε από τους ε, Ιρανούς για να αλλάξει η ε, συμφωνία αυτή, η ρήτρα Sunset, ε, να αναγκάσουμε, να αναγκάσουμε να επιτρέψουν την παρακολούθηση, την επιτήρηση, ε, ας πούμε, των στρατιωτικών βάσεων. Υπάρχουν και μια σειρά από άλλα στοιχεία που πρέπει να αλλάξουν σε αυτή τη συμφωνία που είναι ε, εναντίον μα και πρέπει να, ε, να, να αναγκάσουμε του Ιρανού να αλλάξουν συμφωνία αυτή που του αρέσει τόσο πολύ. ενδεχομένω να το κάνουν αυτό μόνο οι ΗΠΑ. προ τα εκεί κινούνται τώρα. Τώρα δεν πρέπει να βοηθήσει η, η Ευρώπη τις ΗΠΑ αντί να βοηθά το Ιράν να αποκτήσει σε 13 χρόνια πυρηνικό πλουστάσιο Πρέπει να διαρωτηθεί η Ευρώπη. Πού στέκεται η Ευρώπη, πού. Είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτή τη στιγμή πιεστικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κούπερ Βάσα. Ακούσαμε τη φωνή του Ισραήλ. Και τώρα ο κύριος Γκέρετ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Συγχαίρω τον Γιώση. Πέρασε στο στρατιωτικό τομέα την καριέρα του και μόνο τρει διαφάνειε παρόλα αυτά χρησιμοποίησε στην παρουσίασή του. Αυτό είναι επίτευγμα σε αυτού του κύκλου υπηρέτησα στη μυστική υπηρεσία, τη CIA κάποτε. Και δεν θέλουν εκεί οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν διαφάνειε, όπω καταλαβαίνετε. Δεν θα δείξω την παραμικρή διαφάνεια. Πάντα είναι σημαντικό όταν μιλάς για την εξωτερική πολιτική τον είπα στη Μέση Ανατολή ότι πρέπει να τονίσεις τη συνέχιση αυτή, τη συνέχεια που έχει. Δύσκολο σε αυτή τη φάση αυτή η συνέχεια. Διότι είναι πολύ ε, ε, ευμετάβλητη η πολιτική στη Ουάσιγκτον και οι Ριπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί ε, δεν μπορούν να χωνέψουν οι μεν τους δε. Και πρέπει να τονίσει κανείς ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν προβληματίζεται ιδιαίτερα από την ασυνέπειά του, παρόλο που οι ανώτεροι σύμβουλοι του προβληματίζονται. Δύσκολο λοιπόν να περιγράψω επακριβώς την αμερικανική εξωτερική πολιτική για τη Μέση Ανατολή σε αυτή τη φάση, διότι είναι ασαφής η πολιτική και για εκείνους που τη διαμορφώνουν. Πρέπει να πούμε ότι πάντα πρέπει να υπογραμμίσουμε το θέμα της συνέχειας. Αν δείτε στον παρελθόν τι έκανε ο πρόεδρος Ομπάμα, είναι σωστό να πούμε ότι είχε δύο πυλώνες στην προσέγγιση για τη Μέση Ανατολή. Το ένα ήταν η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ο ένας πυλώνας. Ο άλλος πυλώνας και πρώτα η μυστική και μετά η ανοιχτή πυρηνική διπλοπανία με την Ισλαμική Δημοκρατία που οδήγησε στο σχέδιο δράσης και τη συμφωνία με το Ιράν, Ιράν Ιράν-Δίου. Βλέποντας τι κάνει ο πρόεδρος Τραμπ μέχρι τώρα. Και ας πάμε μέχρι τον Ιανουάριο. Ακόμα και φαίνεται σαν αιωνιώτης, ακόμα και να πάμε μόνο πίσω μέχρι τον Ιανουάριο. Η πτυχή της εξίσου που αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας παρέμεινε ίδια. Ακόμα δεν έχουμε εξωτερική πολιτική για τη Μέση Ανατολή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε αντιτρομοκρατική πολιτική για τη ΣΥΠΑ στη Συρία, αντιτρομοκρατική πολιτική για τη ΣΥΠΑ στο Ιράκ, αντιτρομοκρατική πολιτική για τη ΣΥΠΑ στην Ιεμένη και μπορεί να συνεχίσετε σε όλη τη Μέση Ανατολή, αλλά δεν υπάρχει κοινό παρονομαστή όλων των πολιτικών, εκτός του ότι οι ΙΠΑ προσπαθούν να διαλύσουν το Ισλαμικό κράτος ή την Αλκάιδα. Δεν υπάρχει μια μεγάλη ευρία στρατηγική. Ίσως αυτή αναπτυχθεί. Για να συμβεί κάτι τέτοιο θα περιστρέφεται γύρω από ένα θέμα, το Ιράν, αν υπάρξει τέτοια σφαιρική πολιτική. Ίσως ξέρετε κάποιοι από εσά ότι υποτίθεται ότι θα είχαμε μια μεγάλη αναθεώρηση του θέματο του Ιράν. Θα το έκανε αυτό η κυβέρνηση τον Αύγουστο, επισκόπηση τη πολιτική για το Ιράν. Φτάσαμε τέλο Σεπτεμβρίου. Δεν φτάσαμε ακόμα στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Φαντάζομαι ότι ρυθμίζουν τις μικρολεπτομέρειες και θα ανακοινώσουν σύντομα και θα δημοσιεύσουν, υποψιάζομαι, ή θα υπάρξει, θα διαρροή μια και μιλάμε για την Washington, την νέα έκθεση για το Ιράν. Έτσι θα ξέρουμε ποια είναι η πορεία και στρατηγική της κυβέρνησης. Ίσως, ενδεχομένως, να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο οι ΙΠΑ προσεγγίζουν τη Μέση Ανατολή. Από τώρα και στο εξή θα έλεγα, τώρα μα δούμε, αν δείτε τι κάνει η κυβέρνηση Τραμπ στη Συρία και στο Ιράκ, τι βλέπει κανείς. Βλέπει κανείς να διαμορφώνεται μια συνέχεια και αλλαγή. Ο πρόεδρος Τραμπ υπήρξε πιο επιθετικός από ότι ο πρόεδρος Ομπάμα στη Συρία. Απίθανο να είναι λιγότερο επιθετικός από τον πρόεδρο Ομπάμα στη Συρία. Άρα δεν βλέπουμε τεράστια αλλαγή. Δεν βλέπουμε ακόμα κάποια στρατηγική από πλευρά των ΗΠΑ η οποία να, να πιέζει την Ισλαμική Δημοκρατία ούτε στο Ιράκ ούτε σε άλλες περιοχές. Αν δείτε πραγματική πίεση θα τη βλέπατε με μεγαλύτερη χρήση του στατιωτικού δυναμικού των ΗΠΑ, θα αναπτυσσόταν περισσότερα στατεύματα ή θα χρησιμοποιούνταν πιο επιθετικές κυρώσεις. Με πιο επιθετικό τρόπο οι κυρώσεις. Τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβη. Υπάρχουν κάποια σχέδια που κυκλοφόρησαν στο Λευκό Η ΕΠΑ θα ήταν πολύ πιο επιθετική σύμφωνα με τα σχέδια στη Συρία πάνω από 5.000 στρατεύματα της Αμερικής θα ήταν στη Συρία, θα αναπτυσσόταν εκεί, και αντί να υπάρχουν επιθέσεις κατά του Ισλαμικού κράτους, που σχεδόν έχει τηθεί, την επαύριο θα, στόχος θα ήταν η Ισλαμική Δημοκρατία, που τώρα ελέγχει όλα τα στατέματα των Σιητών και των Συρίας και κυριαρχεί και στα υπολείμματα του Συριακού στρατού. Συνέβη κάτι τέτοιο. Από ό,τι βλέπουμε, αντίθετα από το Αφγανιστάν, όπου ο πρόεδρος υποστήριξε τη διατήρηση αμερικανικών δυνάμεων και αύξηση μάλιστα αυτών, μέχρι τώρα, από ό,τι μπορούμε να δούμε, δεν υπάρχει και μεγάλος ενθουσιασμός στο Λευκό Οίκο να γίνει κάτι τέτοιο στη Συρία. Αν με τι άλλο, στο Ιράκ φαίνεται η διάθεση να είναι προ την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή μείωση του αριθμού των στρατευμάτων στο Ιράκ. Περίπου 6.000 στρατεύματα έχουμε. Αυτό έχει δημοσιοποιηθεί. Αυτό ο αριθμό ίσω να είναι μεγαλύτερο από αυτό, αλλά δεν βλέπουμε ακόμα καμία επιθυμία από πλευρά Λευκού Οίκου να αυξήσει σημαντικά την παρουσία των Αμερικανών στο Ιράκ. Κάτι απαραίτητο για να υποστηριχθούν οι Σιήτες που είναι κατά της Ιρανικής επιρροής και να υπάρξει και εμπιστοσύνη στους Σουνίτες ότι δεν πρόκειται να συμφριβούν μετά την κατάρρευση την πλήρη του Ισλαμικού κράτους. Περιμένουμε να συμβεί αυτό. Όλες αυτές οι δράσεις εξαρτώνται από την απόφαση του Πρόεδρου Τραμπ όσον αφορά την περιοχή και τη συμφωνία. Θα ξέρουμε μέχρι Οκτώβριο, 15 Οκτωβρίου τι θα γίνει. Διότι όπως σας είπα, όλα όσα συμβαίνουν στη Ουάσιγκτον ε, διαραίουν πριν ανακοινωθούν. Θα ξέρουμε κατά πόσο ο πρόεδρος αποφασίσει να ακυρώσει τη συμφωνία την πυρηνική με το Ιράν. Αν το κάνει αυτό, πρέπει να θυμηθούμε και σημαντικό ότι δεν θα την ακυρώσει ε, μέσω της συνήθους διαδικασίας, αλλά μέσω νομοθετήματος που περάσει από το Κογκρέσο. Μια πράξη για μια αναθεώρηση της πυρηνικής κατάστασης που κρατεί στο Ιράν και ο Πρόεδρος θα έχει το δικαίωμα να απομακρυνθεί από την συμφωνία για τα πυρηνικά όποτε πιστεύει ότι αυτή η συμφωνία δεν είναι για το καλύτερο δυνατό όφελο των ΗΠΑ. Αν ο πρόεδρος Τραμπ αποφασίσει να την ακυρώσει, γι' αυτό θα το κάνει σίγουρα θα έχει διάφορες υποσημειώσεις όπου θα αναφέρεται σε διάφορα θέματα. Έχουν παράξει περισσότερο βαρύ είδωρο από ό,τι έπρεπε, έχουν περισσότερε μονάδες ε, κεντροφυγικές κλπ. Και ανάπτυξη πυράβλων επίσης. Ε, η ανάπτυξη πυράβλων είναι κάτι που έχει αγνοήσει, ε, όπως η απόφαση 2231 του ΟΗΕ για την ανάπτυξη πυράβλων. Δηλαδή, ποιο είναι το ζουμί, ότι η συμφωνία αυτή κάθε αυτή είναι πολύ κακή ιδέα. Αυτό προωθεί η κυβέρνηση. Κακή ιδέα για τι ΗΠΑ. Αν αυτό συμβεί. Υπάρχουν τρει δυνατότητε, λοιπόν που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πρώτη, ο πρόεδρος επικυρώνει τη συμφωνία. Βλέποντας αυτά που είπε δημοσία, ότι μισεί τη συμφωνία και δεν ήθελε να την κυρώσει τον Απρίλιο και Ιούλιο και το έκανε με κάθε δισταγμό τελικά διότι η ανώτερη συμβουλή του δεν του δίνει τη δυνατότητα να μην την κυρώσει. Άρα εξ αυτού συνεπάγεται ότι ο πρόεδρος τελικά θα ακυρώσει αυτή τη συμφωνία. Συναισθηματικό προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί. Αν την κυρώσει, πιστεύω ότι πιθανότατα ότι η συμφωνία του Ομπάμα θα γίνει η πυρηνική συμφωνία του πρόεδρου Τραμπ. Και δεν θα γίνει άλλη προσπάθεια να διαλυθεί η συμφωνία ή να υπάρξει απομάκρυνση από τη συμφωνία ή να συμπληρωθεί εκτός αν κάνουν κάτι ανόητο οι Ιρανοί και όπως είπε και ο Γιώση πραγματικά αυτό δεν είναι προς συμφέρον του Ιράν να κάνει με τέτοια ανοησία διότι τώρα έχουν μια ομαλή ανεμπόδιστη πορεία προς ουσιαστική πυρηνική υποδομή. Δεύτερη δυνατότητα ο πρόεδρος να αποφασίσει να την κυρώσει αυτή τη συμφωνία και τότε δεν κάνει και πολλά πράγματα. Τι πρέπει να παρακολουθήσουμε σε αυτή την περίπτωση. Είναι τι θα κάνει ο πρόεδρος με τη συμφωνία Boeing. 17,1, 17,2, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο δεκαδικό ψηφίο είναι. Είναι συμφωνία της Boeing, όπου έδωσε άδεια για αυτή τη συμφωνία ο πρόεδρος Ομπάμα και ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να ανακαλέσει αυτή την άδεια. Αν αποφασίσει, α συγγνώμη να κάνω λάθος αν αποφασίσει να καταργήσει τη συμφωνία της Boeing, με το, της Boeing με το Ιράν, αυτό δείχνει σαφώς ότι δεν θα κρατήσει μάλλον το status κουβό να σας πω ότι αν η συμφωνία Boeing καταρρύπτεται και η συμφωνία της Airbus. Είναι αλληλένδετες οι συμφωνίες λόγω περιορισμού ε, όσον αφορά το περιεχόμενο, αμερικανικά ε, ανταλλακτικά και κομμάτια που πηγαίνουν σε κάθε αεροσκάφος Airbus. Άρα θα είναι θέμα ενδιαφέρον για διατλαντικό διάλογο. Η δυνατότητα λοιπόν να παραμείνει το status quo, εκεί αυτό ελπίζουν οι Ιρανοί. Εκτός βέβαια από την κύρωση που αυτό προτιμούν. Υπήρξαν κάποιες δηλώσεις, κυρίως εκείνου που πρέπει να προσέχουμε. Του Αλή Σαλαχή, που είναι ο πρόεδρος του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί στο MIT και έχει πάρει διδακτορικό στην ε, πυρηνική μηχανολογία. Ο Σερέχη πιστεύει λοιπόν ότι οι Αμερικανοί μπορεί τελικά να ε, μην κυρώσουν τη συμφωνία και να επιβάλλουν κάποιες μικροκυρώσεις που δεν θα επηρεάσουν και πάρα πολύ την κατάσταση. Και λίγο πολύ συνεχίζεται το status quo, παρόλο που ο Αμερικανικός Πρόεδρος δεν κυρώνει τη συμφωνία, δεν θα ανταποκριθεί, θα κινηθεί το Κογκρέσο και τελικά δεν θα αναζωπηρωθούν οι γενικές σοβαρές κυρώσεις, μόνο μικρές κυρώσεις θα επιβληθούν που, θα εφαρμ... που μπορούν να γνωρίσουν και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί. Αυτή είναι η δεύτερη δυνατότητα. Η τρίτη. Ο πρόεδρος τελικά δεν κυρώνει τη συμφωνία και τελικά εφαρμόζει αυτά που είπε. Η επιλογή 3 πιθανότατα θα οδηγήσει σε απόσυρση της αδείας που έχει δοθεί στην Boeing και σε ένα κύμα κυρώσεων ε, και τελικά θα, θα ζητηθεί και η διάλυση του, ε, του επαναστατικού σώματος του Ιράν των, των φρουρών της Επανάστασης. Αυτό θα πλήξει την Ιρανική οικονομία, κυρίως στρατηγικούς τομείς της Ιρανικής οικονομίας, ε, που είναι οι τομείς που οι Ευρωπαίοι και οι Ασιάτες ενδιαφέρονται για αυτούς. Διότι εκεί υπάρχει το πολύ, το παραδάκι αυτό θα επηρεάσει άμεσα οι εσδήποτε ευρωπαϊκές και ασιατικές επενδύσεις και θα παγώσει ε, κάθε επένδυση. Δεν θα υπάρξει κάποια ευρωπαϊκή τράπεζα που θα θέλει να εμπλακεί σε κάποια δράση χρηματοδοτική δοθησών των κυρώσεων που θα τους κυνηγούν και των κυρώσεων που κάποιες ευρωπαϊκές ε, τράπεζες ε, πλήρωσαν κατά το παρελθόν. Και τρέμουν τώρα δεν θέλουν να χρηματοδοτήσουν κάποια σημαντικά προγράμματα εντός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Ε, όπως είπα, υπάρχουν διάφορες ε, διαφορές που μπορεί τελικά, διαφοροποιήσει του σχήματος που περιέγραψα και συνδυασμοί. Ο πρόεδρος μπορεί τελικά να προσπαθήσει να κρατήσει συμφωνία ε, της Boeing, να μην κυρώσει την συμφωνία και να επιβάλλει μεγάλες κυρώσεις στο Ιράν. Θα είναι μεγάλος πονοκέφαλος, δεν ξέρω πώς θα συνδυαστούν όλα αυτά αλλά ξέρουμε ότι ασυνεπώς κινείται ο πρόεδρος Τραμπ. Πήγε πρώτα σε εγκαταστάσει στη Νότια Καρολίνα και στις εγκαταστάσεις της Boeing αφού εξελέγει. Δηλαδή τελικά δεν κινείται με κάποια συνέπεια. Δεν πάει προβλέψει, είναι Α, Πιθανότατα λίγο πολύ θα ισχύσει μια από τις επιλογές που είπαμε. Θα κυρώσει, δεν θα κυρώσει και δεν θα κάνει όμως πολλά. Το Κογκρέσο δεν θα κινηθεί δεν θα επιβάλλει ξανά τις παλιές κυρώσεις και δεν θα επιβληθούν κυρίως οικονομικές επώδυνες κυρώσεις ή ο Πρόεδρος τελικά δεν θα κυρώσει και η Boeing θα ακυρωθεί και θα επιβληθούν πολλές ενδιαφέρουσες κυρώσεις με άμεσο αντίκτυπο για πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Αν ο Πρόεδρος ακολουθήσει την τρίτη διαδρομή, ίσως η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ να αλλάξει και σε κάποια άλλη περιοχή, σε κάποια άλλη χώρα της περιοχής. Ίσως άλλη προσέγγιση στη Συρία και στο Ιράκ να ακολουθηθούν. Ενδεχόμενο είναι, δεν γνωρίζω. Υπάρχουν, ε, είναι απρόβλεπτες οι συμπεριφορές του Πρόεδρου. Εξαρτάται θα κάνουν και οι Ιρανοί. Πώς θα αντιδράσουν στην κίνηση του Πρόεδρου. Ένα πράγμα σας εγγυώμαι. Εάν οι στρατιώτες των ΗΠΑ, είτε στο Ιράκ, είτε στη Συρία, οι ειδικέ δυνάμεις, εάν αρχίσουν να πεθαίνουν στα χέρια των Σιητών, τότε θα είναι νεκρή αυτή η συμφωνία. Ε, το Συμβούλιο και ο Πρόεδρος δεν θα ανεχθούν οι Ιρανικές δυνάμεις να σκοτώνουν Αμερικανούς στρατιώτες και ταυτόχρονα να τους, ε, μην τους επιβάλλουν κυρώσεις, εξαιρέσα τις κυρώσεις. Είναι μια αντίφαση αυτή καθε Βέβαια, εξωτερική πολιτική, αμερικανική, όπως όλες οι εξωτερικές πολιτικές, περιέχει αντιφάσεις, αλλά είμαι αρκετά βέβαιος ότι αυτή είναι μια αντίφαση η οποία δεν θα μπορέσει να σταθεί. Αυτό εξαρτάται από το τι θα κάνουν οι Ιρανοί. Η ανταπόκριση του, των Ιρανών θα είναι προσεκτική αρχικά, αν δείτε τις συζητήσεις, πώς το παρουσιάζουν εξωματιούχοι των Ιρανών και υπάρχει πολύ υλικό πάνω σε αυτό. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι λοιπόν πιθανότατα δεν θα κινηθούν ασύμετρα και ασύμετρο στα περσικά σημαίνει το ίδιο όπως τα αγγλικά. Δηλαδή να σκοτώσουν Αμερικανούς στρατιώτες. Δεν προβλέπω να γίνει κάτι τέτοιο στην αρχή. Είναι δυνατόν, είναι απόλυτα δυνατόν, εν συνεχεία, οι Ιρανοί να αντιδράσουν με έναν τρόπο βίο αργότερα. Ίσως να επηρεαστεί και το Ισραήλ. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό τώρα οι Ιρανοί να επιτρέψουν η Χεσμπολά να βομβαρδίσει με πυράβλους το Ισραήλ από τη στιγμή που υπάρχουν λιβανικές δυνάμεις στο Ιράκ και στη Συρία. Δεν νομίζω ότι οι Ιρανοί μπορούν να αφήσουν τη Χεσμπολά να κινηθεί το τρόπος αν επιτόπου στη Συρία αναπτυχθεί η κατάσταση διότι ο τρόπο ή αλλάξει η τακτική και γίνει πιο επιθετικό το Ιράν, ίσω οι Ιρανοί μπορεί να ανάψουν πράσινο φω και να αρχίσουν πάλι βομβαρδισμοί πυραυλικοί σφοδροί κατά των Ισραηλινών. Υπάρχουν και άλλες συνιστώσεις που είναι ενδιαφέρουσες. Το θέμα το κουρδικό, το κουρδικό δημοψήφισμα και αυτό παίζει ρόλο σε σχέση με το τι θα κάνουν οι Αμερικανοί στη Συρία και στο Ιράκ. Τώρα θα λέγω ότι οι Αμερικανοί δεν θα υποστηρίξουν τους Κούρδους στο αίτημά του για ανεξαρτησία. Αυτό μπορεί να αλλάξει. Τώρα, αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια που κινούνται με αυτόν τον τρόπο οι Κούρδοι. Όμως πρέπει να επιληθούν τα γενικότερα ζητήματα. Τι σημαίνει αυτό, ότι οι Αμερικανοί θα, δεν θα χρησιμοποιήσουν σαν βασικό παράγοντα την αντιτρομοκρατία στη διαμόρφωση εξωτερική πολιτική. Η καταπολέμηση τη τρομοκρατία θα μειωθεί σαν παράγον και μεγαλύτερα στατικικά ζητήματα θα αποκτήσουν προτεραιότητα. Η αντιμετώπιση Ισλαμική Δημοκρατία θα διαμορφώσει περισσότερο την Αμερικανική πολιτική και βασικά θα ξέρουμε τα πάντα μέχρι στις 15 Οκτωβρίου όπου, όπως σας είπα, σε μερικές μέρες θα μάθουμε κάτι, διότι φαντάζομαι ότι ο πρόεδρος είπε στο σύμβουλό του για θέματα εθνικής ασφαλείας τι θα κάνει όσον αφορά τη συμφωνία για τα πυρηνικά. Του είπε, φαντάζομαι, τι θα κάνει με τη συμφωνία της Boeing και ο στρατηγός Μακμάστερς γνωρίζει και όλοι οι άλλοι τα αυτά επίπεδα γνωρίζουν. Σε 24-48 ώρες θα έχουμε διαρροή των ειδήσεων. Και μετά μπορούμε να ξανακουβεντιάσουμε για το τι μέλη γενέστε. Αλλά υποψιάζομαι αυτό που σας είπα, επιλογή 1, 2 ή 3 είναι οι μόνες δυνατότητες. Και ίσως να είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι εξελίξεις ανάλογα με το ποια πόρτα θα ανοίξει ε, ο πρόεδρος που θα αφορά βέβαια και τις διατλητικές σχέσεις. Αυτά και σταματώ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι παρουσιάσεις. Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο για τη συζήτηση. Σας παρακαλώ λοιπόν να είστε σύντομοι στις ενδεχόμενες ερωτήσεις. Γιος Ευχαριστώ πολύ. Ήταν δικαίω και το στεφτιστικά όλα αυτά. Αν κοιτάξει κανείς ε, την ε, περίπτωση του Πεκίνου και της Ρωσίας στην αστρολογία. Αν στραφούμε, εδώ βλέπουμε ότι θα μας πούν και αυτοί ότι έχουμε τρεις ε, επιλογές. Αλλά από πού προέρχονται, από πού εξαρτώνται, ποιες είναι οι αντικειμενικές ε, σκέψεις στις οποίες βασίζονται. Στα ζάρια τις έχουμε βρει. Πού, μου φαίνεται να υπάρχει ασυνέπεια. Και πολλές φορές χρησιμοποιείται αυτό. Εγώ νομίζω ότι σε αυτή την περιοχή, αν δει κανείς ε, τις διάφορες καταστάσεις, η ασυνέπεια είναι προφανής. Παραδείγματο χάρη στήριξη αρκινής κυβέρνηση κατά τον ΙΠΑ, που είναι ο καλύτερο φίλο ε, του Ιρανικού καθεστώτος ταυτόχρονα. Δεν ξέρω αυτά που κολλάνε μεταξύ τους, ε, αν θέλω να κάνω κάποιες κριτικές ερωτήσεις. Και το άλλο ερώτημα, Ιδίω σε σχέση με την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν. Το να την ε, καταγγείλουμε, αυτό θα φέρει περισσότερη διαφάνεια και θα είναι πιο προβλέψιμο το Ιράν. Ε, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει κάτι τέτοιο μία συμφωνία νομίζω ότι είναι καλύτερη από καμία συμφωνία. Αυτή είναι η δική μου άποψη και πρέπει να το ξέρει και το Ισραήλ και η Αμερική ότι εμείς μένουμε σε αυτήν την άποψη ότι καλύτερα αυτό από το τίποτα. Είχαμε ακούσει και κάποιε απειλέ από τον κύριο Νετανιάχου και δεν είχαν γίνει συμφωνίε τελευταία. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη μα και τα πολιτι, τις πολιτικές ε, παραμέτρους. Αλλά αυτό το προειδοποιητικό χτύπημα, το preemptive strike, δεν ξέρω. Νομίζω ότι υπάρχουν σημαντικέ υποχρεώσει ε, και διάλογο που πρέπει να γίνεται όχι μόνο με τους εταίρους μας, αλλά και με ε, συνομιλητές όπως είναι το Ιράν. Και για την περίπτωση Βόρειας ακόμη εγώ λέω ότι καλύτερος ο διάλογος ε, παρά αυτός ο φραστικός ε, ριζοσπαστισμός που παρακολουθούμε και είναι κρίμα και από το Βορειοκορεάτη δικτάτορα και από τον Αμερικανό πρόεδρο που κινούνται στα ίδια επίπεδα τελικά. Εγώ καθ' περίμενα κάτι διαφορετικό για έναν εκλεγμένο πρόεδρο σε σχέση με έναν μη εκλεγμένο δικτάτορα αλλά ακολουθούν την ίδια πολιτική. Κύριε Πάσκου, δύο πράγματα. Το πρώτο θα είναι η το αποτέλεσμα της συμφωνίας δεν ήταν επαρκώς σαφές. Ότι δηλαδή ε, θα ενισχυόταν το Ιράν ε, από, να, στις κινήσεις του από τη στιγμή που θα τους είχε δοθεί ε, carte blanche ε, για να κάνουν αυτό που θέλουν ή δεν ήταν σαφές η ιδέα ήταν ότι είναι ένα κόστος που αναλαμβάνουμε και θα το αντιμετωπίσουμε αν προκύψει ή όταν προκύψει. Δεύτερη ερώτηση. Πώς μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει απρόβλεπτο όσον αφορά τα μέτρα απέναντι στο Ιράν από πλευράς Αμερικανικής διοίκησης. Λογικά εγώ θα έλεγα. Δεν, έχει, δεν έχουν αναλυθεί λογικά οι ε, συνέπειες κάθε εναλλακτική και το απρόβλεπτο συνίσταται στο ότι δεν έχει προηγηθεί λογική ανάλυση των συνεπειών. Αν υπήρχε, ε, εγώ θα ήμουν σε θέση να γνωρίζω τις συνέπειες ε, κάποιας πορείας και άρα θα μιλούσα για προβλεψιμότητα. Επειδή ε, συνομιλούμε με λογικούς σε παράγοντες. Και τώρα όσον αφορά τη Βόρεια Κορέα, βλέπω ότι έχει αξία ο διάλογος, συμφωνώ, είναι καλύτερο από οτιδήποτε άλλο. Θα έλεγα ότι πρέπει να υπάρξει αυτοσυγκράτηση κυρίως από πλευράς αυτών που βρίσκονται είναι πιο όριμοι, αλλά διαρωτώμα πώς αντιμετωπίζεις τον άνθρωπο αυτό. Δεν μπορείς να τον αντιμετωπίσεις, δεν μπορείς να τον χειριστείς. Δεν, δεν, δεν γίνεται. Η Κίνα και η Ρωσία λένε, ναι, μην το κάνεις αυτό. Και οι Ηνωμένε Πολιτείες αντί να τους πει κάντε το εσείς όπως νομίζετε ή πείτε μου πώς να το κάνω, δώστε μου ένα αποτέλεσμα, δεν το κάνει αυτό. Δεν το κάνουν αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά τη γνώμη μου υπάρχει και ένα θέμα ότι υποκινούμε τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Κάποιος από πίσω χειρίζεται την κατάσταση. Αυτά. Ευχαριστώ κύριε Βαλέρα. Θα μιλήσω σουηδικά. Εδώ είμαι. Είναι μονομερής η κατάσταση. Έχουμε επικεντρωθεί στο Ιράν και τις ΗΠΑ αλλά πολλοί είναι οι παίκτε στην περιοχή για του οποίου δεν μιλήσαμε πολύ. Χαίρομαι που αναφέρθηκαν τελικά οι Κούρδοι, διότι αποτελούν σημαντικό κομμάτι της προσπάθειας ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή. Πρέπει να δούμε και τις άλλες ομάδες που υπάρχουν εκεί. Και δεν είναι μόνο το θέμα ότι θα γίνει ε, δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία στο Νότιο Κουρδιστάν υπάρχει και το, η δυτική περιοχή του Κουρδιστάν όπου είναι εμπόλεμη αλλά που μπορεί και πάλι να εγκατασταθεί κάποιο είδους δημοκρατία αν τους υποστηρίξουμε παρκώς. Η Τουρκία είχε αντιταχθεί σε αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να λέγατε δύο λόγια περισσότερο από αυτού. Και μετά έχουμε και τη Σαουδική Αραβία Ούτε αυτή αναφέρθηκε πολύ, πέραν του ότι, ότι είναι η καλή. Καθώς διαχωρίζουμε τους μουσουλμάνους σε καλούς και κακούς. Η Σαουδική Αραβία λοιπόν ε, έχει τον πόλεμο με την Ιεμένη Επίσης αγοράζει πολλά όπλα από την Ευρώπη και τις Ηνωμένε Πολιτείες, πράγμα που την κάνει σημαντικό παίκτη στο θέμα της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε δύο λόγια περισσότερο για το ρόλο της Σαουδικής Αραβίας. Εδώ στο Κοινοβούλιο επανειλημμένως έχουμε προτείνει να βάλουμε, να επιβληθεί εμπάργο όπλων Αραβία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Νάρτ. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ να είναι πιο σύντομες οι παρατηρήσεις σας. Ήδη έχουν έρθει οι ομιλητές του επόμενου πάνελ. Μετά τον κύριο Νάρτ, μάλλον θα κλείσουμε τον κατάλογο των ομιλητών, ώστε να δώσουμε τον λόγο σύντομα στους, ε, στα μέλη του πάνελ. Ναι, κύριε Πρόεδρε, αν μιλάμε για τη Μέση Ανατολή. Υπάρχει μια εκοφαντική ε, απουσία των Αράβων που είναι και η πλειοψηφία, πολύ σημαντικός παράγοντας ε, διεθνούς εμβέλειας, είπα και τοπικής εμβέλειας ε, το Ισραήλ, αλλά λείπει η άλλη πλευρά. Μας λένε οι εκτός για τους Άραβες και για τους ουρανού. Ε, θα ήθελα την επόμενη φορά να έχουμε μια ισορροπημένη εκπροσώπηση στο βήμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αντιτρομοκρατία. Από τότε που αποφάσισε το 1808 ο Ναπολέον να... Ε, εισβάλλει στην Ισπανία. Κατάλαβε ε, και καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι χωρίς ε, το λαό δεν γίνεται τίποτα. Έχουμε στο Αφγανιστάν ε, διεφθαρμένα καθιστά το ένα μετά το άλλο τα υποϋποστηρίζουμε. Ο τοπικός πληθυσμός ξέρει και βλέπει τι γίνεται. Βλέπει δηλαδή εμείς να υποστηρίζουμε τους διεφθαρμένους που τους κακομεταχειρίζονται και τους εκμεταλλεύονται και εμείς είμαστε χριστιανοί. Αυτοί μας θεωρούν σταυροφόρους όμως. Εγώ ξέρω το Αφγανιστάν και την, ε, τον πόλεμο εκεί γιατί ήμουν ε, πολεμικός ανταποκριτής και ξέρω γιατί μιλάω τώρα. Για τον Τραμπ και τη Μέση Ανατολή. Ο κύριος ε, Κούπερ Βάσερ είπε ότι είναι ρεαλιστή, συντηρητικός ο Τραμπ, λίγο υπερβολικό όταν έχει ορίσει έναν τελώ αναλφάβητο σε θέματα ε, πολιτικές όπω είναι ο κ. Κούσνερ ε, να είναι μέντορα τη επίλυση των ζητημάτων τη Μέση Ανατολή, ενώ αυτός ε, είναι εντελώ αδαής και το μόνο που ξέρει είναι να κερδοσκοπεί με τα κίνητα. Γιατί βηρητό καλό είναι, αλλά όχι για την επίλυση των προβλημάτων της Μέσης Ανατολή. Και όταν παρατηρούμε τελικά τι έγινε στο, στη Μέση Ανατολή, τι έκανε πρώτον με αυτό το αποτρόπιο καθεστώς ε, των Σαουδαράβων λοιπόν ε, εκεί με αυτούς συμμάχησε και δημιουργεί και τη στρατιωτική βάση, ε, στρατιωτική βάση εκεί και με την Ιορδανία, το ΜΑΝ και τον ε, Κουβέιτ που παρότι έχουν ιδίως το Κουβέιτ πήρε την οικογένεια Σαούντ όταν είχε εξοριστεί το 1800 κτλ είναι ο οχαβιστές και στο Κατάρ και σε Οδική Αραβία, το ίδιο αν θέλετε. Και το τρίτο σημαντικό είναι ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα της Σαουδικής Αραβίας, που εσείς λέτε ότι είναι υποδειγματικοί και συντηρητικοί ρεαλιστές ε, και αυτοί, ε, βλέπουμε ε, τι κάνουν στην πράξη. Και δεν έχει καμία σημασία ότι μέσω της Νταντάουα ε, διαδίδεται ε, η βαχαβητική ιδεολογία. Εμένα μου φαίνεται πραγματικά πάρα πολύ περίεργο που έρχεται να μας κάνει το Ισραήλ μαθήματα για την πυρηνικοποίηση. όταν δημιούργησε ουσιαστικά τη βάση για την πυρηνική βόμβα. Έχετε 100 εσείς και δεν επιτρέπετε πρώτον να μην γίνει λόγος για αποπυρηνικοποίηση της Μέσης Ανατολής και ούτε μιλάτε τι, το παραμικρό δεν λέτε για τις βόμβες που έχετε εσείς. Μην έρχεστε να μας λέτε εσείς και να μας κάνετε μαθήματα εσείς από το Ισραήλ. Δηλαδή να έρχεται ο πολύγαμος να μιλάει για αγαμία. Και έχουμε το ψήφισμα της 25ης Οκτωβρίου 2016. Μπορεί να έχουμε πραγματικά σημαντικές διαφορές με το Ιράν, αλλά υπάρχει κάτι το αποφασιστικό που έχουμε κατάλαβει. Χωρίς τη Σαουδική Αραβία, χωρίς το Ιράν, χωρίς την Τουρκία, χωρίς τη ΣΥΠΑ, χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι δυνατόν να επιληθεί το Μεσαντολικό και να σκεφτόμαστε τώρα ότι θα πρέπει να αφήσουμε εκτός ένα βασικό παίκτη Αλχάσελ Σάμπι, τις ε, λαϊκές πολιτοφυλακές ε, που εμπόδισαν το Ισλαμικό κράτος να μπει στη Βαγδάτη. Δεν μ' αρέσουν και εμένα οι πολιτοφυλακές αυτές, αλλά από τη... Ε, άμα το δούμε πολιτικά και αυτή τη στιγμή, χρειάζονται. Θα είχε μπει το Ισλαμικό κράτος στη Βαγδάτη, αν δεν υπήρχαν. Ούτε εμένα μ' αρέσουν αλλά μου αρέσουν πολύ περισσότερο από το Ισλαμικό κράτος, αν μπορώ να το πω έτσι. Εδώ, όπως είπα, υπάρχει και μια άλλη κφαντική απουσία, Παλαιστίνη, και ένα από τα σημαντικά ε, ζητήματα που υπάρχουν. Ακόμη και ο Βασιλιά τη ορδανία, ο Αμπνταλάχ, που είναι ρεαλιστή, που είναι πραγματιστής, ε, αντιλαμβάνεται ότι δεν ε, μπορούμε να ε, μην λαμβάνουμε υπόψη μας την Παλαιστίνη. Έχουμε τις συμφωνίες ε, του Όσλο. Το Ισραήλ τώρα δημιουργεί ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα, διότι δεν αφήνει να δημιουργηθούν τα δύο κράτη που είναι η μόνη δυνατή λύση. Και βέβαια με τον επικισμό πλέον προοδευτικά αυτό γίνεται αδύνατο. Τι θα κάνετε με τους Παλαιστινίους 50 χρόνια ακόμη κατοχή για να δείτε μπας και εξαφανιστούν από προσώπου γης ενώ προχωρούν οι επικισμοί που παραβιάζουν τις συμφωνίες του Όσλο, αλλά και τον κοινό νου, γιατί απαγορεύουν έτσι την δημιουργία δύο κρατών. Αυτό είναι το θεμελιώδες πρόβλημα που απέ, απουσιάζει εντελώ από αυτή τη συζήτηση. Ούτε εκπρόσωπος από την Παλαιστίνη υπάρχει εδώ. Παρακαλώ λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, επόμενη φορά το πάνελ να είναι πολύ πιο ισορροπημένο. Mr. Mm-hmm. Uh, this panel was called... Ακούστε, κύριε Νάρτα. Κατάσταση Μέση Ανατολή είναι ο τίτλος του θέματος, είπα και Ισραήλ. Αυτό είπαμε, προοπτική είπα Ισραήλ. Αυτό είναι το θέμα. Φυσικά και θα ακούσουμε και άλλες προοπτικές και το κάνουμε συνήθως αυτό. Φυσικά ε, δεν ε, θα μπορέσω τώρα να επιτρέψω ε, να γίνει μια συζήτηση σε σχέση με την πολύ μακροχρόνια ε, μεσανατολική αυτή διαμάχη. Θα παρακαλέσω τους πανελίστες ε, να, αν συμφωνούν, να δώσουν γραπτό υλικό για αυτό το θέμα. Γιατί χρόνο δεν έχουμε πολύ απλά για μια τέτοια συζήτηση. Λυπούμε πολύ. Και τώρα θα δώσω το λόγο για δύο λεπτά στον καθένα από τους ομιλητές μας, γιατί έχουμε ένα Επόμενο κλεισμένο των θηρών, πολύ σημαντικό για την κατάσταση ασφάλειας στη Βόρεια Κορέα. Λυπούμε. Yeah, I know, but I've already... Το ξέρω, αλλά έχω ήδη κλείσει τον κατάλογο. Ναι, λυπάμαι. Είχα σηκώσει το χέρι μου εδώ και μισή ώρα. Σας παρακαλώ να κάνετε μια σύντομη, σύντομη ερώτηση. Δεν πρόκειται να βγάλω λόγο, ναι. Ήθελα απλώς να πω ότι θα συμφωνείτε ίσως όλοι. η πρώτη φορά που είχαμε πρόεδρο ή διοίκηση στις ΗΠΑ που είναι εξίσου απρόβλεπτο, όσο απρόβλεπτος είναι ο παρόν. Ακόμα και αν φτάσουμε πίσω στον ε, στην κρίση των πυράβλων της Κούβας υπήρχαν πάντοτε άνθρωποι γύρω από τον Τζον Κέννεντι που μπορούσαν να μας απαντήσουν τι σκέφτεται. Τώρα δεν μπορεί κανείς να μας πει τι σκέφτεται ο πρόεδρος αν σκέφτεται. Οι ασυνέπειες ε, ε, υπο, υπονομεύουν την κατάσταση. Ο κύριος Κούσνερ αναφέρθηκε ήδη και θέλω να επιστρέψω στη συνάντηση του πρόεδρου Τραμπ με τον κύριο Νετανιάχου πριν λίγες μέρες στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με τον τύπο, το μόνο που συζήτησαν ήταν η ειρηνευτική διαδικασία της Μέσης Ανατολής, αλλά δεν μίλησαν για το Ιράν προς, την, για, προς λύπη του κυρίου Νετανιάχου. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε ακούσει κάτι άλλο σχετικά. Και δεύτερον, ο κύριε Κούμπεβάσορ, μιλήσατε πολύ για το Ιράν και κανείς δεν, ότι κανείς δεν παρακολουθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του. Ποιος παρακολουθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ, δεν ξέρω κανείς ε, να το κάνει αυτό. Και άλλη ερώτηση, γιατί δεν αναφέρατε καθόλου ότι η IDF, η Mossad και η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών του ζητάνε να μην ξανανοίξει η συμφωνία. Υπάρχουν άνθρωποι ειδικοί στον τομέα που έχουν άποψη εντελώ διαφορετική από τη δική σας. Ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στα μέλη του πάνελ. Δυστυχώ ο χρόνος μας είναι πάρα πολύ περιορισμένο. Σα ζητώ να είστε σύντομοι, πολύ σύντομοι. Πρώτο κύριο Κούπερ Πραγματικά θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Ε, η, καμία συμφωνία είναι καλύτερη από μια κακή συμφωνία. Αυτό προσπαθούσα να εξηγήσω. Και γιατί είναι η συμφωνία αυτή κακή. Ενδεχομένω να διαφωνήσετε μαζί μου, εντάξει, αλλά εγώ αυτό που ισχυρίζομαι είναι ότι δεν πρόκειται μόνο για κακή, πρόκειται για φοβερή συμφωνία. Γιατί επιτρέπει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό πλωστάσιο σε λίγα χρόνια. Θα το δούμε αυτό είναι μια πολύ κακή εικόνα. Αυτό μην το ξεχνάμε. Βεβαίω ο διάλογο είναι καλύτερο από την αντιπαράθεση. Κανένα δεν ζητάει αντιπαράθεση, διάλογο ζητάμε, αλλά ο διάλογο να οδηγήσει σε καλή συμφωνία, όχι κακή. Το ίδιο με την Βορεια Κορέα και ο διάλογο εδώ είναι καλύτερο από την αντιπαράθεση. Μερικέ φορέ όμω δυστυχώ ο διάλογο αποτυγχάνει. Αλλά βασικά ο διάλογο είναι καλύτερο από την αντιπαράθεση. Προφανώ ξέραμε σε τι θα οδηγήσει αυτή η συμφωνία. Το ξέραμε και γι' αυτό το είχαμε πει από πριν ότι δεν είναι καλή η συμφωνία. Βγήκαμε από τον δρόμο μας, ασχοληθήκαμε να πούμε ποιες θα είναι οι συνέπειες και οι επιπτώσεις της συμφωνίας. Παρά τα αυτά, η ρευστότητα κάποιων στον, στο, στη Δύση μας οδήγησε σε αυτή τη συμφωνία. Ε, αυτή είναι η πολύ πικρή αλήθεια περιλαμβανομένων και του θέματος της μετανάστευσης στην Ευρώπη, η οποία ξεκίνησε αμέσω, αμέσω, μετά τη συμφωνία. Ξεκίνησε το κύμα ε, μετανάστευση στην Ευρώπη, γιατί στη Μέση Ανατολή, οι οποίοι ήταν κλειδωμένοι μέσα σε αυτό τη διαμάχη πραγματιστές εναντίον ε, ε, ριζοσπαστών, είπαν ότι θα ε, κερδίσουν οι ριζοσπάστε και παρετήθηκαν, έφυγαν. Να δείτε τα στοιχεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το κύμα τη μετανάστευση. Μόνοι σα. μπορείτε να το διαπιστώσετε. Αυτά επ' αυτού. Δεν θα αναφερθώ σε όλα για τους Κούρδους. Κάποιοι αναφέρθηκαν στους Κούρδους. Εσείς νομίζω, ναι δεν είναι το βασικό θέμα στη Μέση Ανατολή. Επηρεάζει τους πάντες, αλλά δεν είναι το βασικό. Δεν είναι η βασική διαφωνία. Επηρεάζουν όμως πολλούς. Οι Κούρδοι έδειξαν ότι είναι αξιόπιστοι και ότι αξίζουν κάποιο είδους ανεξαρτησία. Τώρα, το τι είδους ανεξαρτησία συζητείτε. Αξίζουν την ανεξαρτησία τους. Ε, νομίζω ότι απέδειξαν ότι ε, την αξίζουν οι KOG γιατί έφεραν το μεγαλύτερο βάρος του πολέμου κατά του ISIS και αυτό θα πρέπει να μεταφραστεί σε κάποιο αποτέλεσμα. Η Σαουδική Αραβία και ο ρόλος της. Δεν είναι μόνο η Σαουδική Αραβία, οι πραγματιστές τους οποίους αναφερόμουν στην αρχή έχουν άποψη για το ποια θα πρέπει να είναι η εικόνα της Μέσης Ανατολής. Δεν ε, εμπιστεύονται τους φιλελεύθερους της Δύσης. Δεν τους εμπιστεύονται. Προτιμούν, προτιμούν να συνεργαστούν με εμά, ε, το Ισραήλ, με τους συντηρητικούς της Δύσης που είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν μαζί τους. Και είδαμε πρόσφατα ε, τον τρόπο με τον οποίο η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία και κυρίως τον Μπαχρέιν έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία της Μέσης Ανατολή, ειρηνευτική ε, διαδικασία της Μέσης Ανατολή με το Ισραήλ. Ακόμα και στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ε, υπήρχε μια ένδειξη προς όλους ότι κάτι αλλάζει με αυτούς. Και φαίνεται αυτό και στην αλλαγή κυβέρνηση. Νέα γενιά αναλαμβάνει, η οποία έχει διαφορετική άποψη. Λοιπόν, σας, σας παρακαλώ, τελειώνετε. Ναι, δύο λόγια μόνο για, για το IE hey, το, το Ισραήλ ξέρετε ότι δεν αποτελεί, ε, αποτελεί για κανέναν και παρότι οι Ιρανοί δεν ήταν έντιμοι απέναντι στο MPT και προσπαθούσαν να πάρουν πυρηνικά όπλα για να αλλάξουν τον κόσμο. Είναι κάτι που δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Αντί λοιπόν να καταδιώκουμε το Ισραήλ, θα, είναι, θα έπρεπε να σταματήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι στο οποίο πρέπει να βοηθήσει η Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Γκερέκτ. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ λιτός. Ε, τώρα, η γενική δήλωση σε σχέση με την δίκηση του Ομπάμα, αν ήταν αγαθή ή αν ήταν ε, κάτι άλλο, νομίζω και τα δύο ήταν. Ήταν τα πάντα. Δεν ήθελαν ε, συμφωνία. Πράγματι ισχύει για τον Ομπάμα και τον Τραμπ. Το θέμα είναι πώς είσαι διατεθειμένος να χρησιμοποιήσεις την βία, την ισχύ ε, στον, ε, στην εξίσωση με το Ιράν και τα πυρηνικά όπλα. Στην περίπτωση του Ομπάμα ήταν σαφώς όχι. Και από εκεί προέκυψε η συμφωνία. Δεν γνωρίζουμε εάν ο πρόεδρος Τραμπ είναι διατεθειμένος να χρησιμοποιήσει ε, ισχύ. Ε, αν αν δούμε ποια είναι η κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία, θα πούμε όχι, δεν είναι διατεθειμένος και άρα η λογική είναι ότι ο Τραμπ είναι Ομπάμα υπαριθμών 2. Και αν επανέλθουμε στις αρχικές μου επιλογές, η μεγαλύτερη πιθανότητα υπάρχει για την πιθανότητα ένα από τη δύο και η τρία. Άρα δεν ξέρουμε γιατί ο Τραμπ δεν, δεν προβλέπεται, είναι απρόβλεπτος και είναι δύσκολο να πούμε. Τώρα, όσον αφορά το Κουρδιστάν, είναι λάθος νομίζω ότι ε, ε, εξοπλίζουμε εθνικές ομάδες για να πολεμούν η μία την άλλη. Είναι λάθος ε, των Πολιτειών που χρησιμοποιούμε τους Κούρδους για να απολεμήσουν τους Σύρους. Θέλεις να κάνεις πόλεμο, πας μόνος σου, δεν θέλεις βοηθητικούς και ε, να ε, εξοπλείς άλλους και το σκέλος αυτό του ΠΚΚ είναι στραμμένο κατά της Τουρκίας. Τώρα, όσον αφορά τους Σαουδική Αραβία. Ένα είναι ο βασικό κανόνα στη Μέση Ανατολή ότι η Σαουδική Αραβία που ε, αν κάνουν κάτι θα, το χαλάσουν οπωσδήποτε. Η ιστορία με την Ιεμένη είναι η ουσία ότι θα δημιουργήσουν εκεί και ένα ακόμα κλάδο του, ε, της Χεσμολά. Και επίσης θα πω κάτι, ενδεχομένως να ε, κατηγορούσα, το, μπορώ να κατηγορήσω τον κύριο Κουσνέρ για πολλά, αλλά όχι για τα προβλήματα μεταξύ Κατάρ και ε, Σαουδικής Αραβίας. Και το θέμα του, των πυρηνικών του Ιράν είναι σημαντικό για την Ευρώπη. Το θέμα αυτό στη Βάσινγκτον και για τους δημοκρατές και για τους ρεπουμπλικάνους δεν είναι ε, πολύ σημαντικό. Και ο πρόεδρος Ομπάμα δεν ε, άφησε πολλά περιθώρια και δεν θεωρώ ε, ότι η διοίκηση αυτή θα ασχοληθεί πολύ από αυτό. Ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρος. Ε, ευχαριστώ συνάδελφοι που ήσασταν σύντομοι. Ευχαριστούμε πολύ για το θέμα αυτό της ημερήσιας διάταξης. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τα μέλη του ΠΑΡΕΛ και απευθεία θα περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης και κλεισμένων των θυρών.